Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα σήμερα. Προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε κατευθείαν. Αν δεν υπάρχουν προτάσεις για αλλαγή της ημερήσιας διάταξης, θεωρώ πως εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του Προέδρου, πρώτο θέμα. Έχουμε όλες τις γλώσσες στη διάθεσή μας εκτός όχι μαζί με τα κροατικά. Η μόνη γλώσσα που δεν έχουμε είναι τα αισθονικά. Άρα λοιπόν έχουμε καλή βάση για να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Στις 4 Ιουνίου θα διεξαχθεί μια ακρόαση για τον νέο Κροατή Επίτροπο στις 9.30 μέχρι τις 12.30. Η ακρόαση θα διεξαχθεί σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και όπως συνηθίζετε σε αυτές τις ακροάσεις, το 10% των ερωτήσεων ανήκουν στη δική μας επιτροπή. Και σας καλώ όλους να το χρησιμοποιήσετε. Επίσης, στις 30 Μαΐου έχουμε μια άλλη εκδήλωση για την ασφάλεια των ασθενών στο, στην αίθουσα 1G2 από τις 3 και 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. κύριος Ρώση θα προεδρεύσει, η κυρία Σόμερ, ο κύριος Τέγερ. Μετά στις 18 Ιουνίου, από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, με εισηγητή τον Chris Davis, έχουμε την έκθεση εφαρμογής του CCS. Θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Στις 18 Ιουνίου θα διεξαχθεί μια εκδήλωση για την επισητιστική κρίση θα σας ενημερώσουμε για το που θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου από τις 1 μέχρι τις 2.30 περίπου. Θα διεξαχθεί επίσης μια εκδήλωση για την ανοσοποίηση. Όσον αφορά το τριμερή διάλογο τώρα, έχουμε πολλά να δούμε. Καταρχάς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα μας... Ο κύριος Τόμας Ούλμερ θα συμμετέχει στον τριμερή διάλογο για τα οχήματα, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα οχημάτων στις 3 Ιουνίου. Μετά, breakfast omnibus, τριμερής διάλογος. Ο τριμερής διάλογος διήρκησε περίπου 20-25 λεπτά. Είχαμε πολύ, καλή, πολύ καλό αποτέλεσμα. Προσαρμόσαμε λοιπόν το κανονισμό στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τρίτος τριμερής διάλογος στις 17 Ιουνίου. Για το έβδομο πρόγραμμα δράσης τώρα. Στις 22 Μαΐου. Τώρα, σημείο 3 της μερίσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών για τις 20-21 Μαρτίου, 26 Μαρτίου, 24-25 Απριλίου και 6-7 Μαΐου. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, τότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Μετά προχωρούμε στο σημείο 4. Εδώ έχουμε την πρώτη συζήτηση για την έκθεση ΡΙΣ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο κατευθείαν στην εισηγήτρια. Παρακαλώ, κυρία ΡΙΣ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βασικές γραμμές, γιατί ήδη έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα επανειλημμένως, που επίσης όπως σήμερα θα δούμε μόνο τον επίλογο του, να σας πω ότι είναι οι βασικές γραμμές και οι βασικές συστάσεις ε, για τη δεύτερη ανάγνωση στην οποία συμφωνήσαμε το Συμβούλιο υπέρ ενός νέου κανονισμού για αυτά τα συγκεκριμένα τρόφιμα. 14 Νοεμβρίου του περασμένου χρόνου η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου ολοκλήρωσε τη συμφωνία με το Συμβούλιο. Τότε είχαμε Κυπριακή Προεδρία. Μετά από ένα τελευταίο τριμερή διάλογο που τελείωσε τις μικρές ώρες. Είναι λίγος κόσμος εδώ σήμερα το πρωί, αλλά ήθελα πάντω να σα ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Μίκο, τον κύριο Μαφιουδάκη και τον κύριο Μπορλέ από την Κομισιόν <coughs> για το ενεργό του ρόλο. Δεύτερη σημαντική ημερομηνία ήταν ο Δεκέμβριο του 2012 όπου εκρίναμε το σχέδιο εδώ σε αυτή την Επιτροπή και έπειτα δεύτερη ανάγνωση Απρίλιος 2003. Τώρα, επί τη ουσίας, πιο ενδιαφέρον είναι ότι πετύχαμε τρία βασικά σημεία που απόψε θα τα ψηφίσουμε. Το πεδίο εφαρμογή που θα περιορίζεται στις κατηγορίες πληθυσμού που πραγματικά χρειάζονται αυτά τα ειδικά ε, προϊόντα, τα νεογέννητα, τα παιδιά κάτω των τριών ετών, τους παχύσαρκους, ε, και τους ασθενείς που είναι ε, αυτή τη στιγμή ε, σε ε, στα νοσοκομεία, αλλά και τα παιδιά που γεννιούνται με χαμηλότερο βάρος του κανονικού, του μέσου όρου. Ε, όλες, όλα τα υπόλοιπα διατροφικά προϊόντα, όπως δημήτριακά, σνακ κτλ, θα μεταφερθούν για την ώρα στην νομοθεσία General Food Law. Τώρα, οι δυσανεξίες τύπου λακτόζης και γλουτένης που ήταν σημαντικές στη διάρκεια της συζήτησης, ήταν μια από τις προτεραιότητες που εκφράστηκαν στη διάρκεια της συζήτησης, ενσωματώνονται

στον κανονισμό για την ενημέρωση προς τους καταναλωτέ, ε, που είναι προσφυλή στην κυρία Σόμαρ και που προβλέπει παρόμοιους κανόνες για τις αλλεργίες. Ε, ε, πιστεύω πως απάντησα στον κύριο Ρώση γιατί εισήγαγε τροπολογίες, κατέθεσε τροπολογίες τελευταία στιγμή. Δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή αλλά ελπίζω πως θα τον δω το απόγευμα στην ψηφοφορία γιατί οι ανησυχίες του φυσικά και καλύπτονται από τις συμβιβαστικές μας προτάσεις. Να υπογραμμίσουμε τη σημαντική νίκη στον τομέα της σήμανσης γιατί πείσαμε τα κρατημένα μελη να επεκτείνουν ε, τους περιορισμούς σήμασης, ας πούμε για τις φωτογραφίες μωρών, για τα μωρά από 6 μέχρι 12 μήνες ήταν ε, ένα ιδιαίτερο αίτημα της κυρίας Σαρμπού από τους σοσιαλιστές που όλοι υποστηρίξαμε. Επίσης υπογραμμίζω την διαρκή ανησυχία της Επιτροπής μας για διαγραφή των ε, νανοσωματιδίων, νανοηλικών Ε, και επίσης απαγορεύονται τα φυτοφάρμακα, αυτά που θεωρούνται ως ε, ενδοκρινικοί διαταράκτες. Η Κομισιόν διευκρινίζει στην ε, δήλωσή της που προσαρτάται στη συμφωνία να συνεχίσει τον αγώνα για να περιορίσει την ύπαρξη κίνδυνων φυτοφαρμάκων ε, στα τρόφιμα και πολύ συγκεκριμένα στα ε, εν λόγω τρόφιμα. Καλό λοιπόν την Επιτροπή να επιβεβαιώσει την ψηφοφορία του 2012 και να στηρίξει αυτή τη συμφωνία που είναι εξαιρετική, την οποία συνάψαμε με το Συμβούλιο και που θυμίζω απερίφθησαν να περίψουμε τις έξι ε, τη, τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα ΕΕΦΤΕ. Να ευχαριστήσω τους σκιώδες που είναι παρόντες και τους υπόλοιπους. Ε, μίλησα για την κυρία Δελάν και την κυρία Ζαρμπού, τον κύριο Σλούτερ και βεβαίως να ευχαριστήσω. Ξέρω πως δεν είναι επίσημη η διαδικασία, αλλά ήταν σημαντική η βοήθεια ε, της γραμματείας ε, που μας στήριξε μέχρι τέλος, ε, κυρία Όλιγκερ, Σαλάσκη, και να θυμίσω πως το μήνυμά μας είναι απλό στην ουσία, ότι δηλαδή τα βρέφη και τα, α, α, οι, σοβαρά ασθενείς δεν είναι καταναλωτές όπως όλοι οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χρύς. Οι ισχυώδεις εισηγητές τώρα θα λάβουν το λόγο. Η κυρία Ντελάνγκη έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Έχουμε κάνει το, το έργο μας. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτό το νομοθέτημα στην αρχή σε μια πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Αυτή ήταν και η συμφωνία που κάναμε. Ίσως οι εκπρόσωποι της Κομισιόν θα ήταν πρόσφορο να λάβουν το λόγο και να υπενθυμίσουν τη συμφωνία που πετύχαμε για την γλουτένη όπου εδώ αυτό το, το θέμα καλύπτεται όχι με ειδική νομοθεσία, αλλά μέσω του νομοθετήματος για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Αλλά για τους ασθενείς ή για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα, τίποτα δεν θα αλλάξει. Έχουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για το θέμα αυτό, ώστε στην πράξη να μην αλλάξει τίποτα, <clears throat> παρά το γεγονός ότι η τα τρόφιμα με γλουτέν για άτομα που έχουν δυσανεξία δεν θα βρίσκονται σε ένα ειδικό πλαίσιο, αλλά θα είναι μέσα στα πλαίσιο της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές. Γνωρίζω ότι θα υπάρχουν τροπολογίες από την ομάδα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για το θέμα αυτό, αλλά η γλουτένη ήταν ένα από τα κέρια ζητήματα που συζητήσαμε σε όλες τις συνεδριάσεις που κάναμε με το Συμβούλιο. Ας μην ανατρέψουμε λοιπόν τη συμφωνία για αυτό το λόγο γιατί νομίζω ότι η συμφωνία καλύπτει και τα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να σας πει περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο κύριος Πούλη για την ε, Κομισιόν έχει το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Non, à ce stade, je voudrais... Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα κυρίω να ευχαριστήσω την κυρία Ρίστη, την εισηγήτρια και του σκιώδει εισηγητέ για τον ενθουσιασμό με τον οποίο ασχολήθηκαν με αυτήν την πρόταση που κάναμε. Είναι μια φιλόδοξη πρόταση. Αλλάξαμε τελείω την προηγούμενη ε, νομοθεσία, διατηρώντα τα σημαντικά στοιχεία, όπω είπε και η κυρία Ρή, για τα πιο ευάλωτα άτομα, δηλαδή για τα παιδιά και τα βρέφια και για του ε, αρρώστους. Ε, να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το πρόβλημα της ε, γλουτένης ε, το έχουμε εντοπίσει βεβαίως. Ήταν ένα σημείο συζήτησης ε, αρκετά έντονης και αναλάβαμε την δέσμευση ότι θα το ρυθμίσουμε αυτό στο στην κανονισμό για τη σήμαση Food Information for the Consumer με κατεξιοδότηση πράξης όπου θα ε, φροντίσουμε ώστε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το gluten free και very low gluten. Ε, πάντως δεν θέλω να προτρέξω τις αποψινήσεις της ψηφοφορίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εν γέννη στην Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία και Θέλω να θα σας θέσει ένα ερώτημα. Απλώ να καθησυχάσω την Κομισιόν ότι εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με τις προτάσεις της Κομισιόν. Η ομάδα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας απλώς έθεσε ορισμένες τροπολογίες, αλλά από τη δική μας πλευρά εμείς υποστηρίζουμε απόλυτα τη συμβαστική λύση και δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αρχή της συζήτησης. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΕΕ σήμερα. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ρης. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, λέει η κυρία Ρης. Μια χαρά είναι. Θα δούμε το απόγευμα στη ψηφοφορία τι θα γίνει. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Η ψηφοφορία είναι σήμερα το απόγευμα στις 3 η ώρα. Ωραία, οπότε έχουμε κλείσει αυτό το θέμα και ερχόμαστε στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με εισηγήτρια την κυρία Ροτ Μπέρεντ και η κυρία Ροτ Μπέρεντ είναι υπεύθυνη για το χαρτοβασίλειο που έχουμε μπροστά μας τις πάρα πολλές τροπολογίες που υπάρχουν στο σημείο αυτό και μετά έχουμε και την έκθεση Λίζε πάλι για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά. Παρακαλώ κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, δεν φταίω εγώ που έχουμε τόσο πολύ χαρτί, διότι οι τροπολογίες μου είναι μικρές και ταπεινές. 45. Δεν είναι πολλές, αλλά έχουμε 760 τροπολογίες από τους υπόλοιπους συναδέλφους για την έκθεση αυτή και αυτό δείχνει και πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση. Ε, από τις 8 μέχρι τώρα είχαμε συνεδρία των σχεδόν εισηγητών. Ε, τους ευχαριστώ πολύ που ήταν όλοι παρόντες. Διότι είναι νωρίς για να γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα. Βλέπω ότι δύο είναι εδώ. Και οι υπόλοιποι θα έρθουν σύντομα, βρίσκονταν στην άλλη άκρη του κτηρίου. Θέλω σύντομα να πω ότι Έχουμε τρία σημεία τα οποία είναι αρκετά αμφιλεγόμενα και αυτό φαίνεται και από το πόσες τροπολογίες έχουν υποβληθεί γι' αυτά. Πρώτον, η πρόσβαση στην αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όπως γνωρίζετε, στο κείμενό μου προβλέπω μια κεντρική και μια αποκεντρωμένη ε, διαδικασία έγκρισης διάθεση στην αγορά. Συμφωνούν ορισμένοι συνάδελφοι με αυτό, άλλοι όμως όχι. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα συμβιβαστούμε και μεταξύ μας και με την Επιτροπή, διότι η ασφάλεια των ασθενών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και πρέπει να φροντίσουμε να διατίθενται στην αγορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία έχουν εξεταστεί λεπτομερών. Γνωρίζετε ότι αυτές οι συσκευές ε, δεν παρουσιάζουν δυσκολία στην ε, ανάκτηση κλινικών δεδομένων αλλά και οι μελέτε συχνηλασιμότητας είναι αρκετά περίπλοκε και δύσκολε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί. Κοίταξα αν μπορούμε να κάνουμε μια, ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τη τάξη 3. Ορισμένοι συνάδελφοι συμπεριλαμβάνουν και προϊόντα τη ταξη 2 2β, προϊόντα τα οποία εμφυτεύονται και παραμένουν στο σώμα ή τα οποία περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες ή προϊόντα τα οποία δεν εμφυτεύονται, αλλά εισάγονται στο σώμα με μη μορφή. και διοχετεύουν ενεργές ουσίες στον οργανισμό. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Δεν γνωρίζω αν θα το καταφέρουμε προς το παρόν, διότι έχουμε ακούσει τα πάντα από το να παραμείνει το σύστημα ως έχει μέχρι το να αλλάξει. Είμαι όμως αισιόδοξη πως τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε και μεταξύ μας και με την Επιτροπή. Και σκοπεύουμε αυτό να το κάνουμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτή την έκθεση θα συναντηθούν ή στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή στην αρχή της επόμενης. Έτσι λοιπόν ενδεχομένως την επόμενη Τετάρτη να γίνει και άλλη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Επίσης, Πρόεδρε, όσον αφορά την επανεπερξεργασία, έχουμε και πάλι πολλές τροπολογίες. Εδώ παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει όλα τα προϊόντα που αυτοί χάνουν επανεπεξεργασίας ε, να μεταφέρεται η ευθύνη στους επανεπεξεργαστές και όχι στους κατασκευαστές. Και πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα προϊόντα μίας χρήσης και στα προϊόντα που μπορούν να επανεπεξεργαστούν και τα προϊόντα μίας χρήσης πρέπει να είναι μίας χρήσης. Εγώ προτείνω αυτό να το τονίσουμε, να δώσουμε σαφήνεια στον ορισμό τι είναι ένα προϊόν μίας χρήσης και να παραμείνει ένα προϊόν ε, ως μίας χρήσης εάν, αποδειχθεί, εάν δεν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι δηλαδή μπορεί να επεξεργαστεί, αν δεν αποδειχθεί επιστημονικά. Επίσης, έχουμε πολλές τροπολογίες, όχι μόνο από, τους, από έναν αλλά από όλους, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ορισμένες δεν τις καταλαβαίνω, είναι από την αλήθεια, εκείνες που αφορούν την, ε, τον ορισμό μίας χρήσης. και άλλες επίσης που αφορούν τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά. προτάθηκε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος προϊόντων που είναι κατάλληλα για επανάχρηση. Και τέλος έχουμε το θέμα των κοινοποιημένων οργανισμών τις σελίδες 18 έως 49 έχουμε τις τροπολογίες 481 533. Όλες αυτές είναι τροπολογίες από τους σκιώδεις εισηγητές. Και να σας πω ότι μόνο οι σκιώδεις εισηγητές κατέθεσαν τροπολογίες. Εδώ. Μετά. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μια κοινή γραμμή ότι δηλαδή οι κοινοποιημένοι οργανισμοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με περισσότερη προσοχή. Δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που προτείνω εγώ. Πιστεύω όμως, σε κάθε περίπτωση, ότι οι προϋποθέσεις και η ποιότητα των κοινοποιημένων οργανισμών θα διαφέρει κατά πολύ από το έργο που θα αναλάβουν εάν τους επιτραπεί να κοινοποιούν τα προϊόντα όλων των τάξεων, παρά μόνο των τάξεων 1 και 2α. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να δούμε πώς μπορούμε να συμβιβαστούμε. Ιδανικά, για μένα, εάν δεν υπάρχει έγκριση κεντρική είτε αποκεντρωμένη, ελπίζω να γίνει αλλά δεν είμαι σίγουρη, στην περίπτωση αυτή πραγματικά θα πρέπει να ενισχυθεί η ποιότητα των κοινοποιημένων αυτών οργανισμών. Και πιστεύω πως αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν εσωτερικό προσωπικό, ιατρούς, φαρμακολόγους που να εργάζονται εκεί, ειδικού δηλαδή, Και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται outsourcing. για αυτή τη διαδικασία έγκρισης. Και σε περίπτωση που αυτό χρειάζεται πρέπει να είναι σαφέστατο το ποιος θα αναλάβει αυτή την έγκριση, ποιος εξωτερικός συνεργάτης. Τώρα, όσον αφορά τον μηχανισμό αξιολόγησης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας και εγώ έχω καταθέσει τροπολογίες σχετικές με αυτό. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε είναι τα τρία σημαντικότερα και πιο αμφιλεγόμενα σημεία. Ο μηχανισμός λοιπόν εξέταση, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί και η διάθεση στην αγορά και η πρόσβαση στην αγορά. Ελπίζω πραγματικά να καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε συμβιβασμό γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Είμαι έτοιμη να το κάνω, καλή την πίστη. Ωστόσο, να πω ταυτόχρονα ότι η υποχρέωσή μας είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών. Είναι μια υποχρέωση όχι μόνο για τους ιατρούς, αλλά και για τους... Ε, αλλά και κάτι που περιμένουν από εμάς και οι οργανισμοί των ασθενών και σε αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κλινικές δοκιμές. Ο μηχανισμός της αγοράς και πραγματικά να σας πω ότι δεν έχουμε πολύ περιθώριο για συμβιβασμούς, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το έχω συζητήσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν αλλάξει η πρότασή της για την πρόσβαση στην αγορά, θα μπορούν να μας στηρίξουν. Και θα ήθελα εδώ να ρωτήσω την Επιτροπή, εάν μπορείτε να φανταστείτε κάποια διαφορετική πρόσβαση στην αγορά για ορισμένες τάξεις προϊόντων, για τη 2Β για παράδειγμα. Κύριε Πρόεδρε, δεν με έχετε διακόψει μέχρι τώρα. Είστε πολύ γενναιόδωρος. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Με χαρά μου τώρα να ακούσω τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ναι. Μία φορά μόνο πνίξαμε την εισηγήτρια και δεν την αφήσαμε να συνεχίσει. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο από την προηγούμενη έκθεση που ήταν σύντομη, γι' αυτό λοιπόν τώρα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Προσοχή όμως να παραμείνουμε στο χρονοδιάγραμμά μας. Διότι μετά θα συζητήσουμε την έκθεση του κύριου Λίζε. Αρχίσουμε τώρα με τους σκιώδεις συζητητέ. Προτείνω όλοι να τηρήσετε ένα όριο 4 λεπτών. Κύριε Μακίνες, πρώτη έχετε το λόγο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κάναμε μία <clears throat> συνεδρίαση προγευματική, αλλά χωρίς πρόγευμα για τα θέματα αυτά. Ήταν πάρα πολύ καρποφόρα αυτή η συνεδρίαση, αλλά νηστική Και τελικά πήρα, <laughs> πήρα πρωινό ερχόμενη στη συνεδρίαση αυτή, οπότε δεν είχα πρόβλημα ασυτείας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια για αυτά που είπε και να σταθώ σε μερικά από τα σχόλιά της. Πράγματι λειτουργούμε καλή την πίστη όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το φάκελο. Έχουμε θέσει την ασφάλεια των ασθενών στον πυρήνα της εργασίας μας και ξέρουμε ποιες είναι οι πιέσει σε σχέση με την ε, διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο για συμβαστικέ λύσει. Σε ορισμένε περιοχέ που είναι δύσκολη αυτή η συμβαστική λύση, αλλά μπορούμε να την πετύχουμε. Θα πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή μα και η προγευματική μα στρατηγική ήταν η πιο αποτελεσματική γιατί είπαμε θα αντιμετωπίσουμε λεπτομεριακά όλα τα τεχνικά θέματα και μετά σε πολιτικό επίπεδο <clears throat> θα σταθούμε σε θέματα που είναι σίγουρα πολύ πολύπλοκα. Αλλά το να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα στους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για κοινοποίηση, για καλύτερη ποιότητα προσωπικού, για καλύτερο έλεγχο. Όλα αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά και εγώ θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το θέμα της ε, Παρακολούθηση μετά από τη θέση σε εμπορία και την αναφορά επεισοδίων και προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν. Όλα αυτά είναι τεχνικά θέματα που πρέπει να επεξεργαστούμε και εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Κομισιόν για όλα αυτά τα θέματα τα οποία έθιξε η συγγετρία. Και σας δίνω τον υπόλοιπο μου χρόνο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα σήμερα. Ο κύριος Χόλεν Κάμερ για την Άλντε έχει το λόγο. Είναι γενναιόδωρο το να έχω σήμερα τέσσερα λεπτά. Αυτό δεν συμβαίνει κάθε φορά. Αν δούμε τις τροπολογίες, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο γενικές ε, ομάδες ε, θεμάτων για τα οποία μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Καταρχήν για το ποιε θα πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για τους φορείς κοινοποίηση που θα πρέπει να επιβάλλουμε και νομίζω ότι από τις πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί υπάρχει κοινό έδαφος για συμβαστική λύση πρέπει να προσέξουμε να μην φτάσουμε σε πολύ λεπτομεριακό επίπεδο. Γιατί εμείς ως Επιτροπή δεν μπορούμε να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι είναι λυσιτελές να θέσουμε σαν προϋπόθεση ότι οι ε, εμπειρογνώμονες οι οποίοι προέρχονται από ένα φορέα να μπορούν να ε, παίξουν αυτό το ρόλο, ότι δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά να υπάρχει ένα ειδικευμένο, ένας ειδικευμένο φορέα κοινοποίηση, αλλά να, μπορεί να, ε, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ευρισκόμενοι εντό ενό φορέα εμπειρογνώμονε ήδη. Δεν πρέπει να χάσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του. Και φυσικά μπορεί να υπάρξει και μια ανταλλαγή ε, μεταξύ των φορέων αυτών και των πανεπιστημίων στην πράξη. Ε, δεν είναι λοιπόν ρεαλιστικό να τους αποκλείσουμε από τη διαδικασία αυτή. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προϊόντα που βρίσκονται ήδη στην αγορά. Την ε, παρακολούθηση και την λασιμότητα στα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να βρούμε έδαφος για συμβαστικές λύσεις και συμφωνούμε καταρχήν ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ πιο συχνοί και πιο αυστηροί έλεγχοι από τους ε, παραγωγούς των προϊόντων. Εκεί είναι ο τομέας όπου πολλές φορές μπορούν να υπάρχουν καταχρηστικές ενέργειες, ακόμα και εγκληματικές ενέργειες και πρέπει να προωθήσουμε και την κεντρική διαδικασία έγκρισης. Εγώ ε, λυπάμαι που η συζήτηση έχει γίνει όχι σε επίπεδο ουσιαστικών επιχειρημάτων, σε επίπεδο πεπιθήσεως σε σχέση με το αν πρέπει να είναι κεντρική ή όχι η διαδικασία. Και εάν υπάρξει μια, ένα πρόβλημα με κάποιο φαρμακευτικό ε, σκεύασμα, όπως έγινε με τα εμφυτεύματα στήθους στην Γαλλία, όλα αυτά τα θέματα είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε καλύτερα. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Γαλλίας υπήρξαν υποψίες και για εγκληματικές ενέργειες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κάποια απάτη δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό γιατί η δυνατότητα απάτης υπάρχει και στον οργανισμό κοινοποίησης και με την κεντρική ε, διαδικασία έγκρισης. Δεν μπορούμε απλώς να λύσουμε το πρόβλημα αυτό με το να θεσπίσουμε μια κεντρική αρχή έγκρισης Απλώς θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και να αυξήσουμε τις απαιτήσει ποιότητας αυτού του συστήματος και δεν πρέπει να να ξεχάσουμε το ότι πολλές, πολλά προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με, την, με τον κατασκευαστή ενός φαρμακευτικού συσκευάσματος, αλλά περισσότερο με τη χρήση του συσκευάσματος, παραδείγματος χάρη με την ε, χρήση που κάνουν οι ιατροί αυτών των φαρμάκων. Και τέλος, για το θέμα της ε, μοναδικής χρήσης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορούμε να λύσουμε Πρέπει κάπου να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή τη συζήτηση. Αυτοί οι οποίοι παράγουν ένα προϊόν το οποίο στη συνέχεια ε, δίδεται για επανεπεξεργασία και περνάει μια επανεπεξεργασία στη συνέχεια, ο καθένας σε αυτή την αλυσίδα πρέπει να έχει την ευθύνη για τα θέματα αυτά. Αυτός ο οποίος παράγει αρχικά το προϊόν θα πρέπει να διατηρήσει την ευθύνη για αυτά τα οποία υπόσχεται καταρχήν το προϊόν. Και αυτό ισχύει και για τον επανεπεξεργαστή. Δεν μπορούμε φυσικά να θεωρήσουμε ότι είναι υπεύθυνο ένας παραγωγός ε, φάρμακος για το γεγονό ότι ένα νοσοκομείο χάρη επανεπεξεργάζεται ένα σκεύασμα. Θα πρέπει όμω να έχουμε τι ίδιε ακριβώ απαιτήσει όπω και στον παραγωγό και σε αυτόν ο οποίο κάνει την επανεπεξεργασία. Το αν τώρα θα υπάρχει το θέμα της μοναδικής χρήσης ή όχι, τελικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι θέμα κρίσης και πεποίθησης και δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με απόλυτα ορθολογικό τρόπο. Και ευχαριστώ λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάσει στη διαδικασία συμβαστικών λύσεων. Κυρία Φαρμέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Έρχομαι, ήμουνα στη Μασαλία όπως ξέρετε και έγινε αυτή η δίκη της υπόθεσης ΠΥΠΕ που παρατίθεται εδώ και που μετά αντιποτέλεσε αντικείμενο ψηφίσματος και μετά μας οδήγησε να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την οδηγία. Υπήρχε 5.500 ε, ε, γυναίκες παρούσες ε, που ακριβώς είχαν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της προσθήκης στήθους που είχαν βάλει σιλικόνη βιομηχανική. Τι θα κάνουμε λοιπόν με βάση αυτό το σύστημα που υπάρχει ε, ε, ας το ελέγξουμε. Αυτό το εμφύτευμα είχε επιστοποιηθεί από έναν ε, οργανισμό πιστοποίησης που ήταν γερμανικός. Αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης. Έκαναν ελέγχους και όταν έκαναν τους ελέγχους δεν είδαν τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν είναι απόλυτη εγγύηση για την ασφάλεια των ασθενών. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι όταν η Food and Administration στην Αμερική, η FDA, ζητά έγκριση για εμπορία. Όταν ήρθε και έκανε έλεγχο στην Μασαλία, έμεινε εκεί ένα μία εβδομάδα και είπαν όχι δεν εγκρίνουμε αυτά τα εφητεύματα. Αυτό σημαίνει πως όταν υπάρχει ένας οργανισμός σαν την FDA που έρχεται και ζητά έγκριση εμπορίας και που θα ελέγξει, εκείνοι λένε όχι. Εκεί όπου υπήρξε το πρόβλημα μετά ήταν ότι ξανά έστειλαν το ντοσχέ σε γαλλικό εθνικό οργανισμό που δεν απήντησε στον συναγερμό στην προειδοποίηση της FDA. Τι λέμε λοιπόν ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους. Γιατί εγώ θεωρώ πως οι οργανισμοί πιστοποίησης με όλους τους εμπειρογνώμονες που έχουν Πώς θέλετε να είναι αντικειμενικοί όταν ξέρετε ότι 100% της χρηματοδότησής τους προέρχεται από τους κατασκευαστές. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται από έναν οργανισμό δημόσιο. να κάνουν εκείνη τον έλεγχο, πολύ ωραία, αλλά δεν αρκεί. Η απόδειξη είναι ότι όταν ήρθαν να κάνουν τον έλεγχο του ΠΙΠ δεν είδαν την απάτη, ενώ αν είχαν δει τους λογαριασμούς αυτής της εταιρείας θα είχαν δει ότι υπήρχε πρόβλημα ανάμεσα στη βιολογική, ή φυσιολογική σιλικόνη που είχε λάβει την έγκριση και το νούμερο των φυτευμάτων. Δεν αντιστοιχούσαν αυτά τα δύο. Με, με εντυπωσιάζει λοιπόν ότι για, μιλάμε για ασφάλεια των ε, στενών, ενώ αυτή τη στιγμή οι βιομήχανοι δεν πάβουν να κάνουν απάτες. τελευταία απάτη ήταν ε, το εμφύτευμα Σεραβέρ που είχε γίνει από κάποιον κατασκευαστή και ούτε καν είχαν περάσει από οργανισμό πιστοποίησης και είχαν χρησιμοποιήσει παρόλα αυτά την ε, σήμαση ε, ε, ε, της κοινότητας και πήραν τα νοσοκομεία και κλινικές αυτά τα εφητεύματα και τα τοποθέτησαν σε ασθενείς. Οι βιομηχανοί, αυτοί οι κατασκευαστές είναι που κάνουν τις απάτες και κάθε φορά βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι οι οργανισμοί επιστοποίησης δεν είναι εγγύηση για τους ασθενείς. Και γι' αυτό και έχουμε την εντύπωση ότι για όσα είναι εμφυτεύματα, δηλαδή όσα μπαίνουν μέσα στο σώμα, θα πρέπει να υπάρξει έγκριση, αδειοδότηση για την κυκλοφορία του προϊόντος. Και όταν υπάρχουν επικίνδυνα εμφυτεύματα, ποιος την πληρώνει μετά. Δεν είναι οργανισμοί πιστοποίησης, είναι ο φορολογούμενος που πληρώνει την ύφη και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν οι αδειοδοτήσεις, να γίνονται κλινικές δοκιμές προηγούμενα και όταν μου λένε ναι, αλλά αυτό κάνουν τους ε, κατασκευαστές να χάνουν χρόνο. Ε, ας χάσουν δύο, τρεις, τέσσερις μήνες. Τι αντιπροσωπεύει αυτό σε σχέση με την ζημιά που παθαίνουν οι άρρωστοι από τη στιγμή που πρέπει να τους αφαιρέσουν τις, ε, τα εμφυτεύματα. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι με τη δίκη θα έπαβαν οι απάτες. Ε, όχι λοιπόν. Καθημερινά γίνονται απάτε. Και εγώ δεν εμπιστεύω αυτού του οργανισμού πιστοποίηση που λένε ότι είμαστε καλύτεροι ενώ το 100% τη χρηματοδότησή του προέρχεται από του βιομήχανου. Ε, υπάρχει πρόβλημα λοιπόν στον έλεγχο και υπάρχει πρόβλημα για την εγγύηση τη ασφάλεια των ασθενών. Και όλα τα θύματα, γιατί πολύ θα ήθελα να δείτε τα θύματα στη Μασαλία, όλα τα θύματα ζητούν την ε, ε, αδειοδότηση για την εμπορία. Μπορεί να υπάρχουν δύο επίπεδα, εντάξει, για τα εφητεύματα, για όλα αυτά που είναι επικίνδυνα. Και γιατί όχι και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως κάνει η FDA στην Αμερική. Και ό,τι είναι λιγότερο προβληματικές κατηγορίες να είναι οι, εθνικές, ε, οι εθνικοί οργανισμοί. Αλλά πραγματικά χρειάζονται έλεγχοι για να αγγίθουμε την ασφάλεια των ασθενών. Ευχαριστώ πολύ. Μα είναι για να κουβάκι, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά, έχουμε υποχρέωση να φροντίζουμε την ασφάλεια των ασθενών και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό και θα λειτουργεί ομαλά και δεν θα καθυστερεί την αφροντίδα των που χρειάζονται ασθενείς. Στην συνάντηση των σχεδόν εισηγητών συνειδητοποίησαμε ότι θα υπάρχουν συμβιβασμοί. Το θέμα είναι πού. Αυτό είναι το ενδιαφέρον πώς θα συμβαστεί κάθε ομάδα, διότι το θέμα είναι αρκετά τεχνικό και πιστεύω πως πραγματικά πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με την τεχνητή άποψη και με, ε, τεχνική άποψη και μετά να συζητήσουμε πολιτικά. Σίγουρα οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, το κεντρικό σύστημα, η προέγκριση πριν την κυκλοφορία στην αγορά είναι νευραλγικά σημεία. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι. Όμως να πω ότι όταν Κάνουμε λίγο για απάτη. Εδώ χρειάζονται συστήματα ιχνηλάσιμα. Να ξέρουμε δηλαδή από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ευθύνη η οποία να είναι αναλογική του μεγέθους της απάτης. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να βρούμε κάποιο συμβασμό για το καλό των ασθενών. Ευχαριστώ πολύ. Άλλε όσα επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κυρία Ντάγμα Ροτμπέρεντ έχει ήδη παρουσιάσει την κατάσταση που προήλθε από τη συνεδρίαση των σχεδόν συγητών σήμερα το πρωί, εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα από τα σημεία που αναφέρθηκαν. Δεν νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποφύγουμε να υπάρχει απάτη. Οποιαδήποτε νομοθεσία και αν εγκρίνουμε δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε απόλυτα. Ούτε με αυτή τη ρύθμιση ούτε με άλλη ρύθμιση θα μπορέσουμε ακόμα και με ένα αστυνομικό κράτος δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο να, με το να λέμε ότι θέλουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές ε, Αυτά που είπε η Ντάγμαρ και ο Μισελ τόνισαν τη σημασία της πιστοποίησης και της διαδικασίας έγκρισης προτού τεθεί ένα προϊόν στην αγορά, ένα ιατροτεχνικό προϊόν και φυσικά συμφωνώ και με αυτά που είπε Ντάγμαρ ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου ή αυτά τα οποία αποτελούν αντικείμενο καινοτομία θα πρέπει να έχουν μία έγκριση από ένα κεντρικού χαρακτήρα οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα προϊόντα μπορούν να περνάνε τη διαδικασία έγκρισης σε εθνικό επίπεδο. Μία από τις τροπολογίες που έχει καταθέσει η ομάδα μου πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ε, ανταποκρίνεται σε αυτά που είπε η κυρία Ριβαζή. Όλοι οι εμπειρογνώμονες που κάνουν αυτόν τον έλεγχο, αυτή την αξιολόγηση, θα πρέπει να είναι ελεύθεροι συγκρούσεων συμφερόντων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εγγύηση ότι οι φορείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουν την έγκριση δεν υπόκειται σε συγκρούσεις συμφερόντων και αυτό είναι απαραίτητο για να μην είναι εύκολη της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Πιστεύω επίση ότι η διαδικασία έγκρισης και ο εκ των υστέρων έλεγχος μετά τη θέση σε αγορά είναι τα βασικά στοιχεία του συστήματος. Θα πρέπει να υπάρξει υψηλή ποιότητα και στους ε, φορείς κοινοποίηση και συγχρόνως θα πρέπει να μειώσουμε και να καταργήσουμε η δυνατό τις ε, ατέλειες που υπάρχουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Αυτό είναι απαραίτητο για τους ε, ασθενείς και τους χρήστες αυτών των ιατροτεχνικών προϊόντων. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια νομοθεσία η οποία αντιμετωπίζει από μία πλευρά το επιθυμητό σε επίπεδο καινοτομία, αλλά δεν θέτει ένα αμφιβόλο συγχρόνως την ε, ασφάλεια των ασθενών. Αν τα πράγματα πάνε στραβά δεν θα είναι δυνατό εκ των υστέρων να λύσουμε τα προβλήματα αυτά και να δώσουμε θεραπείες. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής εγγύηση σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση και με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο προτού όλα αυτά τα προϊόντα φτάσουν στην αγορά. Και πιστεύω ότι στις επόμενες συνεδριάσεις μας θα έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα σημεία αυτά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σωστό νομοθέτημα στο τέλος. Ευχαριστώ, όλοι ο Πρόεδρος. Οι υπόλοιποι ομιλητές τώρα. Η κυρία Κούκοβιτς, Μίλαν Κάβανοφ, Ρόσμπαχ, Λίζε. Ξέχασα κάποιον. Ο Ρίχα Επίσης. Η κυρία Κούκοβιτς πρώτη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Γιατί ολοκλήρωσαν ένα πολύ δύσκολο έργο πρέπει να σας πω και έχω καταθέσει επίσης κάποιες ε, τροπολογίες και υποστηρίζω και κάποιες τροπολογίες της συναδέλφου Μαγκίνες, των συναδέλφων Μαγκίνες και Ρόσπαχ. Επλά ήθελα να τονίσω κάποια σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούν νάνο υλικά που μπορούν να απελευθερωθούν στο ανθρώπινο σώμα και αυτή, η, αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να υπόκεινται σε, στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης και στις ίδιες προδιαγραφές συμμόρφωσης, ποιότητας, ασφάλειας ε, όλα λοιπόν θα πρέπει να γίνονται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις ίδιες. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να εκθέσουμε τις ε, γενικές υποχρεώσεις των διαφόρων ε, οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τις μεγάλες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οι οποίες ειδικεύονται στις σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς γιατί είναι πάντοτε δύσκολο κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης για μια μικρομεσαία επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά. Επίσης για, τις, ε, για τα προϊόντα υψηλού κινδύνου <coughs> Προ όφελο τη αυξημένης διαφάνειας, οι κατασκευαστές θα πρέπει να ενημερώνουν τους εμπειρογνώμονες ασφάλειας και διαφάνειας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια, διότι εκεί όπου έχουν διαπιστωθεί περιστατικά θα πρέπει να γίνονται έρευνες για την ασφάλεια. Η, Ένωση, η οδηγία της Ένωσης ορίζει το θέμα της ε, τοποθέτησης στην αγορά και της διάθεσης στην αγορά. Ε, πιστεύω πως θα πρέπει όλοι να συμμορφούνται άμεσα με την ε, οδηγία πριν τοποθετηθούν στην αγορά, διατεθούν στην αγορά, άσχετα εάν πρόκειται για, άμεση, για προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα είτε θα, ή που θα αποθηκευτούν. Και ένα σώμα κοινοποιημένο θα πρέπει να μπορεί να προβαίνει στο έργο του ελέγχου. Η διαδικασία επίσης θα πρέπει να παρακολουθείτε ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο κύριος Κάμπανοχ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν αναφερθεί ακόμα εδώ. Θα ήθελα να, καταρχήν να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη δουλειά που έγινε, για τη λεπτομερή και ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση. Μιλάμε για ένα κανονισμό μια νομοθεσία, ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα πρέπει να είναι σταθερό και προβλέψιμο. Συζητάμε για μείωση ε, των ε, εξουσιών της, των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά την κατεξουσιοδότηση της συμπράξεις. δηλαδή. Εγώ καλωσορίζω την ε, υποχρεώσει για τον κατασκευαστή και τον διανομέα των προϊόντων αυτών. Αλλά δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να διατηρήσει, να Επιβαρύνονται επίσης οι απαιτήσει γλώσσας για την τεκμηρίωση θα πρέπει να απλοποιείται όταν αυτή προορίζεται για διοικητικούς σκοπούς και δεν έχει στόχο τους χρήστες, τους ε, ασθενείς. Άρα δηλαδή δεν δίνει επιπλέον πληροφορίες αυτούς. Τώρα όσον αφορά την επανεπεξεργασία την εκ νέου χρήση επηρεάζομαι πολύ από την προσωπική μου εμπειρία. Θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιοι κανόνες ώστε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη ε, προστασία για τους ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα δεν θα δημιουργούμε εμπόδια ε, στους ε, γιατρούς. Πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρχει ένας αρνητικός ε, κατάλογος ε, ε, συσκευών μίας χρήσης ή προϊόντων μίας χρήσης. Τώρα βέβαια ακόμα και όταν είναι μίας χρήσης πολλές φορές ξανααποστηρώνεται και ξαναχρησιμοποιείται. Έλεγχε και συμμόρφωση προς τους κανόνες. Θέλουμε να έχουμε σαφείς ε, κανόνες ε, ώστε να μπορούν όλοι να τους ε, ακολουθούν και να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό σώμα που θα υποπτεύει την, την, την εφαρμογή των κανόνων. Αλλά εδώ εγώ δεν θέλω να μιλήσω για την επιτυχία ή την αποτυχία των συστημάτων υποπτίας εφόσον κάποιος σαφώς παραβαίνει ξεκάθαρους κανόνες και νομοθεσία. Δεν πιστεύω ότι αν αλλάξουμε το σύστημα χρηματοδότησης θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα είναι σαν να λέμε ότι αυτοί που κλέβουν, οι κλέφτες, αν και απαγορεύεται και η αστυνομία εξασφαλίζει ότι ο κόσμος δεν θα, δεν θα κλέβει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιοι κλέφτες συνεχίσουν αυτή τη δουλειά, η, δουλειά, η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της. Κύριε Ρόσμπαχ, παρακαλώ. Πολλά προϊόντα, για παράδειγμα τα ε, υγρά προϊόντα, παρουσιάζουν πρόβλημα όσον αφορά τη μία χρήση της ε, πολλαπλές χρήσεις. Και όταν ρωτάω τους κατασκευαστές, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι τα προϊόντα μία χρήση είναι σχεδιασμένα για μία χρήση. Και το πρόβλημα όταν χρησιμοποιούνται ξανά είναι ότι πολλές ε, φορές δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι έχουν καθαριστεί σωστά. Γι' αυτό λοιπόν εγώ Είμαι υπέρ της απόλυτης απαγόρευσης επαναχρησιμοποίησης προϊόντων μίας χρήσης. Υπάρχουν ορισμένα προϊόντα βέβαια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από μία φορά, όμως και κάποια άλλα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποστηρωθούν και δεν είναι ασφαλής η χρήση τους πάνω από μία φορά. Εάν όμως δεν μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία κάποια τέτοια απαγόρευση, το κύριο μέλημά μας πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι η ασφάλεια του ασθενούς. Προσωπικά δεν θα επιθυμούσα να χρησιμοποιηθούν πάνω μου τέτοια προϊόντα μια χρήση που έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά. Και πιστεύω πραγματικά πω οι, κατα... ασθενεί έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται γι' αυτό. Όλοι μα εδώ πέρα είμαστε δυνάμοι ασθενεί και όλοι έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε εάν αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά ή όχι. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους ανεξάρτητα από το ποιος χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν μιας χρήσης. Είτε αυτό είναι κάποιος ε, ιδιωτικός επαγγελματίας υγείας είτε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Χρειάζεται επαρκής πληροφόρηση. Και επίσης στηρίζω όλες τις προτάσεις που υποστηρίζουν την ενίσχυση των εμπειρογνωμόνων και των αρμοδιοτήτων του στους κοινοποιημένους οργανισμούς. Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη πιστοποίηση και εντάξει, ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σου έκθεση. Και να πω ότι ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε καλές συμβαστικές τροπολογίες, διότι διαφορετικά ένα θεός ξέρει τι μπορεί να γίνει. Καλή τύχη λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ροτ Μπέρεντ για την πολύ και καλή δουλειά της. Η έκθεσή της συνδέεται άμεσα με τη δική μου, με τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν είναι προς το συμφέρον μας να εναρμονίσουμε τις δύο αυτές εκθέσεις και να έχουμε κοινά σημεία αφετηρίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος και μιας ε, διαδικασίας προέγκρισης. Το είπα και την τελευταία φορά, θα το επαναλάβω για να το διευκρινίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στην τελευταία συνεδρίαση είπα πως είμαι της άποψης ότι μία κεντρική έγκριση θα διαρκέσει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχουμε ένα τελείω καινούριο σύστημα, για παράδειγμα τον, ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αυτή η δημιουργία είναι Ηράκλειο έργο. Πρέπει να βρούμε τους εμπειρογνώμονες που θα επανδρώσουν αυτούς τους κοινοποιημένου οργανισμούς και πιστεύω πως μόνο αυτό έχει ως αποτέλεσμα τεράστιο διοικητικό φόρτο. Τρία χρόνια που προβλέπει η Κομισιόν δεν επαρκούν, πιστεύω. Πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα, αλλά πρέπει να βελτιωθεί γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν και για, άλλα, για άλλους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε στο ισχύον σύστημα και να το βελτιώσουμε. Προσωπικά πιστεύω ότι οι τροπολογίες της Dagmar για, την, για τα προσόντα των ε, υπαλλήλων στους κοινοποιημένους οργανισμούς, είναι προς την, πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης Γράφει στην ε, έκθεση ότι οι εμπειρογνώμονε των ε, κοινοποιημένων οργανισμών πρέπει να έχουν την απαραίτητη εμπειρία, αλλά όλες οι προδιαγραφές είναι κάπως ασαφείς πιστεύω. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πραγματικά τις ε, τροπολογίες τη Εντάγμαρ και στις δύο εκθέσει, και στη δική μου και τη δική τη και να προσπαθήσουμε βάσει αυτέ να βρούμε συμβιβασμού. Επίση, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες και στην δική μου έκθεση και στην δική της, οι οποίες είναι αρκετά αμφιλεγόμενες και αφορούν την ε, αρχή της επικουρικότητας και την ε, τήρησή της. Όσον αφορά τις ε, κλινικές δοκιμές που θα τις ψηφίσουμε το απόγευμα, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μπορούν να απαγορεύσουν την κυκλοφορία ε, στην δική τους αγορά ενός προϊόντος το οποίο θεωρείται ως υψηλού κινδύνου. Όμως πιστεύω ότι εάν ένα προϊόν έχει απαγορευτεί σε μία χώρα δεν πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε άλλες. Ευχαριστώ πολύ Πίτερ Ρεμπέκα Τάιλερ, επόμενη μιλήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να πω σύντομα τα σχόλιά μου για την ε, συζήτηση αυτή. Ε, ήθελα απλά να τονίσω ότι τα θέματα είναι αλληλένδετα και κάποια θέματα που θα αναφέρω για την IVD ισχύουν και για, τις ε, ιατρικούς, ε, για τα ιατρικά, τεχνολογικά προϊόντα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ε, οι οργανισμοί δεδομένων, οι οργανισμοί κοινοποίησης κτλ. Ελπίζω ότι θα τα λάβει υπόψη της η Κομισιόν γιατί πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες οι δύο κανονισμοί. Σύντομα λοιπόν για την πρόταση για τους, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα κύρια στοιχεία ε, της κεντρικής πρότασης της, για την συγκέντρωση της διαδικασίας. Εγώ εξακολουθώ πιστεύω πως ε, τα πλοενεκτήματα μιας ε, τέτοιας διαδικασίας δεν είναι αρκετά για να εισαχθεί και κάτι τέτοιο θα σημαίνει πολύ μεγάλους οικονομικά, οικονομικά οικονομικές δαπάνες και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει εμπειρογνωμοσύνη για, τέτοιους, ε, για τέτοια ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όπως σας είπα τα ουσιαστικά μου σχόλια θα τα διατηρήσω για την συζήτηση περί IVD. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρίχαρτ Ζάμπερ τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πιστεύω πως πρέπει να διατηρήσουμε τα πλεονεκτήματα του υφισταμένου συστήματος της γρήγορης πρόσβασης στην αγορά, όμως να κοιτάξουμε και πώς θα μειώσουμε την γραφειοκρατία. Η δική μου τροπολογία 598 ασχολείται με αυτό και αναφέρει τη δημιουργία ενός νέου άρθρου του 44α το οποίο θα ε, προβλέπει μια υπηρεσία κεντρική, εθνική, εγκρίσεις και εδώ αναφέρομαι κυρίως στα προϊόντα της τάξης 3. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυτή η προτινόμενη κεντρική διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης που προτείνει η Συγκητέ και η Κομισιόν θα είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Και δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στους ε, ασθενείς. Και δεν βλέπω κάποια μακροπρόθεσμα ωφέλη λοιπόν σε αυτό. Καταρχάς πιστεύω πως αυτές οι εθνικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν κοινά κριτήρια και πρέπει επίσης να εμπνέουν εμπιστοσύνη διότι στην τελική ανάλυση αυτές θα εκδίδουν τις εγκρίσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια στο ποιες ουσίες θα υπάγονται και ποια προϊόντα θα υπάγονται στην κατηγορία 3. Πιστεύω όμως πως καλό θα ήταν, όπως πρότειναν και πολλοί συνάδελφοι εξάλλου, να κοιτάξουμε το πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι ασθενείς με τις εθνικές, ε, τους εθνικούς κοινοποιημένους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Και τώρα η Κομισιόν. Ναι. Αν δεν, με, αν σας ενοχλεί κυρία Πρόεδρε, η Σαμπίνα είναι εδώ, αλλά, αλλά θα ήθελα να λάβω το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο και που δίνετε γενικά στην Κομισιόν το λόγο. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και και βλέποντας τον πλούτο και την πολυπικιλία των απόψεων που έχουν καταθέσει οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, είναι πάρα πολύ θετικά αυτά. Εμείς έχουμε κάθε σεβασμό για αυτή την άσκηση και το αίσθημα κατεπήγοντος με το οποίο η εισηγητρία και η Επιτροπή σας αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό και θέλουμε να το προωθήσουμε και θέλουμε να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματα που παραμένουν του του λεχθέντος. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων για τα θέματα της ε, <clears throat> έγκρισης. Δυσκολεύει κάπως το εγχείρημα αυτό, <clears throat> αλλά πόσα έχουμε ακούσει σήμερα είναι σίγουρο κάτι και είναι ένας κοινό στόχος, ένας κοινό ε, στόχος προς επίτευξη είναι η επίτευξη του υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας για τους ασθενείς στην Ευρώπη και θα πρέπει να δούμε όλοι με ποιο τρόπο μπορούμε για τα ιατροτεχνικά προϊόντα να εξασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια σε μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εμπιστοσύνης. Η Κομισιόν γνωρίζει απόλυτα το καθήκον της για τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι θα εργαστείτε αυτή τη βδομάδα σε τεχνικό επίπεδο και θέλω να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε στις συζητήσεις σας στο βαθμό που μπορούμε. Αυτό που έχουμε καταγράψει και στις συζητήσεις αυτές και βλέποντας και τις τροπολογίες είναι ότι η ιδέα μιας απόλυτα κεντρικής διαδικασίας έγκρισης δεν είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει πλήρως την θέση της Κομισιόν η έκθεση αντικτύπου ήδη επεσήμανε το γεγονός ότι αυτό από μόνο του δεν πρόκειται να αυξήσει την ασφάλεια των ασθενών. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει το κοινό σημείο ότι η ενίσχυση των κριτηρίων για τους φορείς κοινοποίηση είναι ένα σημαντικός τρόπος για να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Έχουμε λοιπόν καθήκον να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ασθενών γιατί αυτό είναι η προτεραιότητά μας και είναι επίσης το καθήκον μας να μάθουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος που ανέφεραν πολλοί βουλευτές εδώ. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο ερώτημα της εισηγήτριας, για την επανεπεξεργασία που είναι το άλλο σημαντικό θέμα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόταση της Κομισιόν, η οποία θέτει τον επανεπεξεργαστή στην ίδια θέση από έποψη ευθύνη όπως τον αρχηγό παρασκευαστή, είναι υπαγορευόμενοι από ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης και την αυστηρότητα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι εδώ μπορούμε να βελτιώσουμε όμως αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα νοσοκομεία. Ε, κατονώ αυτό το οποίο είπαν <clears throat> οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Έχουμε ένα καθήκον έναντι των ασθενών που δεν έχουν κανένα έλεγχο για όλα αυτά τα θέματα και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για μια επικοδομητική λύση που θα επιτρέψει και στην Επιτροπή σας να καταλήξει στις 10 Ιουλίου σε μια επικοδομητική ψηφοφορία. Και για να σεβαστώ το χρόνο στο ίδιο πλαίσιο για άλλες τροπολογίες που έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την παρακολούθηση των φορέων κοινοποίησης, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το πλεονέκτημα το οποίο προκύπτει και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για άλλες πολύ επικοδομητικές τροπολογίες όπως το ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης ε, συσκευών ιατροτεχνικού χαρακτήρα που πηγαίνουν τροπολογίες προς τη σωστή κατεύθυνση Βλέπουμε λοιπόν πολλά θετικά στοιχεία εδώ και χαιρόμαστε για τον κατεπήγοντα τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα προτεραιότητα για την Κομισιόν. Θέλουμε να εγκριθεί, συγγνώμη, εγκριθεί στην τρέχουσα νομοθετική περίοδο και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε για τι προσπάθειέ σα, ιδίω τη εισηγητρία. Είμαστε στη διάθεσή σα να σα βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και η εισηγήτρια και πάλι έχει το λόγο για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στη συζήτηση. Με όλες τις τροπολογίες που έχουμε ενώπιόν μας, η συζήτηση έχει φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τα σχόλια των συναδέλφων. Κάποια από αυτά ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Κάποια άλλα σχόλια δεν ακολουθούν απόλυτα τη δική μου γραμμή. Γι' αυτό όμως πρέπει να πρόβουμε και στις συμβαστικές λύσεις. Θέλω απλώς να διασαφηνίσω τα εξής. Δεν θέλω να πέσουμε στην παγίδα που προσπαθούν να στήσουν οι παραγωγοί ιατροτεχνικών προϊόντων. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι οποιοδήποτε άλλο σύστημα θα παρατείνει τη διάρκεια της ε, διαδικασίας έγκρισης και θα δυσκολέψει την είσοδο στην αγορά των προϊόντων αυτών. Ένας οργανισμός παραγωγών με τρομερό, τρομερά συγκινητικό τρόπο μας περιέγραψε την περίπτωση μιας ασθενούς που δεν μπορούσε να πάρει ένα προϊόν που της ήταν απαραίτητο. Εμείς θέλουμε να σταθούμε στην πραγματικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι πρώτες της Κομισιόν που εξετάζουμε ε, αναφέρεται σε ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή θα καλύψει ένα χρονικό διάστημα 7 μηνών, αν πολύ σωστά το βλέπω. Η δική μου διαδικασία προσθέτει μόνο δύο μήνες. Αυτό δεν είναι τίποτα αγαπητοί συνάδελφοι, απολύτως τίποτα. Αν δείτε συγχρόνως ότι οι 7 μήνες που προτείνει δεν σημαίνουν και άμεση πρόσβαση στην αγορά, γιατί στα περισσότερα εθνικά κράτη θα πρέπει να ξεκινήσουν ε, και διαπραγματεύσουμε με τους φορείς κοινωνικής ασφάλειας, ασφάλιση συγγνώμη, που θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα αυτών των προϊόντων και αυτό δεν γίνεται πάντα εν παραλίλω, μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Αν δείτε λοιπόν για τα προϊόντα αυτά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία περνάνε από κεντρική διαδικασία έγκρισης, χρειάζονται πολύ λιγότερο χρόνο για να υπάρξει έγκριση και για την ε, απόδοση κόστους από τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης. Μην δεχτείτε λοιπόν να σας λένε ότι οι νέες διαδικασίες κάνουν λιγότερο ανταγωνιστική την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθυστερούν την είσοδο στην αγορά, όπως λένε τα λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών. Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρόσβαση των ασθενών στα προϊόντα αυτά, αλλά επίσης οι εταιρείε οι οποίες παράγουν αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να το πράττουν αυτό με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ανταγωνιστικός και θετικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ο κύριος Κράμερ ότι δεν υπάρχουν λογικά επιχειρήματα αλλά απλώς συζητούμε σε επίπεδο πεπιθήσεων. Πρέπει να σας πω σαφώς όταν ήρθε η πρόταση της Κομισιόν, εγώ τόνισα ότι δεν είχε καμία σχέση με το σκάνδαλο ΠΙΠ των ευθυνταυμάτων στήθους. Όπως θυμόσαστε, μία πρώην συνάδελφος, η κυρία Μαριωρή, Μαλιώρη, είχε, είχε ζητήσει από την Κομισιόν να προωθήσει κατεπηγόντως την πρόταση αυτή. Υπήρξε λοιπόν αυτό το σκάνδαλο, αλλά αυτό δεν προκάλεσε την πρόταση τη Κομισιόν. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν εγκληματικέ ενέργειε στον τομέα αυτό, εγώ θα σας έλεγα παρόλα αυτά ότι μια κατάσταση πραγμάτων <clears throat> με την διαδικασία αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν, είναι, δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πραγματικότητα αυτή η διαδικασία. Αυτό θα το λέγαμε ούτω ή άλλω και η κυρία Κράμερ δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο. Είναι κάτι το οποίο έλκεται εκ των πραγμάτων. Και φυσικά δεν μπορεί ο κάθε φορέας να έχει στη διάθεσή του τους εμπειρογνώμονες που χρειάζεται. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τους οργανισμούς κοινοποίηση να περνάνε προϊόντα της κατηγορίας 2β, 3 ή ακόμα και 2α με το να ζητούν από κάποιον υπεργολάβο να κάνει την απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Αν θέλετε να το κάνουμε έτσι, θα πρέπει να το κάνουμε και με τα φαρμακευτικά σκευάσματα στο τέλος. Είπε ο κ. Κράμερ χωρίς μικρόφωνο ότι εγώ δεν είμαι δίκαια σε αυτά που λέω και δεν παρουσιάζω την πλήρη εικόνα. Όχι, όχι, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω. Δεν θέλω να είμαι άδικη σε κανένα. Ποτέ δεν το κάνω αυτό. Είπατε ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα αντικειμενικά. Επί της ουσίας είπατε ότι υπάρχουν μονάχα αυτά τα οποία πιστεύει ο καθένας και χρειάστηκε να απαντήσω εδώ, να αντιδράσω. Νομίζω ότι είναι εμπεριστατωμένα τα επιχειρήματα τα οποία σας παρουσιάζω και όχι μονάχα αυτό το οποίο πιστεύω εγώ. Και όταν μιλάτε για τους ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν μόνοι την ευθύνη για τα εμφυτεύματα, είναι γεγονός ότι η επιτυχία ενός εμφυτεύματος μπορεί να συνδέεται και με τον τρόπο ζωής ενός ασθενούς. Αλλά ο ασθενής δεν μπορεί να λάβει όλη την ευθύνη για ένα προϊόν. Αν δείξετε σε ένα ασθενή παραδείγματος χάρη τρία ή τέσσερα διαφορετικά εμφυτεύματα λεκάνης, δεν είναι σε θέση να αποφασίσει. Ακόμα και ο πιο μορφωμένος ασθενής δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αν δείξετε όμως σε ένα ασθενή τα διάφορα αυτά προϊόντα για εμφυτέματα γονάτου ή λεκάνης ή στήθους ή οτιδήποτε, ο ασθενής συνήθως ακολουθεί τη γνώμη του, του γιατρού. Δεν μπορεί να γνωρίζει ο ίδιος. Όπως είπε όμως και ο κύριος Κράμερ, η χνηλασιμότητα είναι ένα σημαντικό σημείο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα καλύτερο σύστημα χνηλασιμότητας για να γνωρίζουμε ποιος έχει κάνει μία εμφύτευση, σε ποιο νοσοκομείο κτλ. Γιατί ένα προϊόν μπορεί να είναι μια χαρά, αλλά ίσως μπορεί ο ιατρός ο οποίος έχει κάνει την χρήση αυτού του προϊόντος να μην, είναι, να μην έχει κάνει σωστά αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ορθοπαιδικούς παραδείγματο χάρη. Και για αυτούς που είπαν ότι πρέπει να εξετάσουμε την επανεπεξεργασία. Εδώ υπάρχουν κάποιες προτάσεις τροπολογιών και από την ανερόσπαχα. Επίση υπάρχουν αυτέ τι προτάσει. Νομίζω πρέπει να επαξεργαστούμε όλα αυτά τα σημεία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Η κυρία Μακίνε έκανε σαφέ από την αρχή ότι υπάρχει πάντα περιθώριο για συμβιβασμού, ότι δεν απέχουν απόλυτα οι απόψει μα, αλλά για κάποια άλλα θέματα είναι δύσκολο να το πετύχουμε και πρέπει να τα επανεξετάσουμε. <clears throat> Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θα προτιμούσα να μην μπούμε σε μια αμφιλεγόμενη διαδικασία ψηφοφορίας για θέματα που είναι ουσιαστικού χαρακτήρα και η Κομισιόν νομίζω ότι μας είπε ότι σε κάποιους τομείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Από τη δική μου λοιπόν απόψη και όχι μονάχα για τα θέματα διαδικασίας, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Αν υπάρξει υποστήριξη μπορούμε να έχουμε μια συνενετική ψηφοφορία αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω δεδομένο επειδή είναι ένα σημαντικό θέμα. Δεν θα ήθελα να καταλήξουμε σε μια ψηφοφορία που απλώς θα εξαρτηθεί από ευκαιριακή πλειοψηφία. Θα ήθελα να βρεθεί μια λύση η οποία βρίσκει όλους σύμφωνους στην Επιτροπή μας και θα μπορούσαμε μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του 2014 να κλείσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ πολύ Στις 10 Ιουλίου θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή εδώ στην Επιτροπή και ενδεικτικά προβλέπεται να πάει το θέμα στην Ολομελία το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση και τις συνεισφορές σας. Τώρα πάμε στην επόμενη έκθεση του Πέτερ Λίζα για τα in vitro διαγνωστικά τεχνολογικό προϊόντα που συνδέεται και με την προηγούμενη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε να ευχαριστήσω καταρχάς τους και εισηγητές για την καλή συνεργασία. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές μέχρι τώρα και πιστεύω πως όλοι μάθαμε ο ένας από τον άλλο και καταφέραμε να βελτιώσουμε την διατύπωση. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία εγώ ίδιος πρότεινα μετά από συζητήσεις με τους σκιώδες εισηγητές και με πυρογνώμονες. Το ένα σημείο το, το ανέφερα ήδη, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει υψηλές απαιτήσει για την ασφάλεια. Για παράδειγμα, ε, πανεπιστημιακή μελέτη συν δύο χρόνια πρακτικής εμπειρίας για το προσωπικό αυτό που θα επανδρώσει λοιπόν τους οργανισμούς αυτούς. Σε ορισμένα δεν υπάρχει προσωπικό που να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις μέχρι τώρα ε, και στα κρατη που υπάρχει Οι απαιτήσει λοιπόν είναι ίδιες και για αυτούς που έχουν και για αυτούς που δεν έχουν. Πιστεύω πως καταρχάς πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση σε αυτό το σημείο προτού δημιουργηθούν ακόμα υψηλότερες απαιτήσει που δεν μπορούν να εκπληρωθούν από όλους. πιστεύω πως η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιγράφει όσο καλά θα έπρεπε τα προσόντα των υπαλλήλων των κοινοποιημένων αυτών οργανισμών. Δεν γίνεται εκείνοι που ελέγχουν τους κοινοποιημένους οργανισμούς να έχουν λιγότερα προσόντα από όσους εργάζονται σε αυτούς τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες για το badge testing όπως λέγεται, δηλαδή για τον τακτικό έλεγχο ενός ε, διαγνωστικού προϊόντος της τάξης 4, της τάξης D. Εδώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε με πολλούς τρόπους το σημείο αυτό και μόνο στις ε, δοκιμές υψηλού κινδύνου παρατηρείται αυτό το πρόβλημα, της τάξης D. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες και δικές μου και συναδέλφων, οι οποίες αφορούν το σύστημα πιστοποίησης. Τα φαρμακεία, για παράδειγμα, και τους διανομής, Εδώ χρειάζεται ένα σύστημα εχνηλασιμότητας, ιδιαίτερα προς αποφυγή ε, πλαστών προϊόντων και χρειάζεται αυτό το σύστημα να είναι ενιαίο. Να υπάρχει δηλαδή για παράδειγμα ένας ενιαίος σαρωτής και όχι πολύ διαφορετική. Τώρα όσον αφορά την ε, συμβουλευτική έχουμε βελτιώσει εδώ την διατύπωση. Πιστεύω πως η συζήτηση ήταν πάρα πολύ καλή και μας οδήγησε σε αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στον ε, τομέα της γενετικής. Εδώ μπορούσαμε να θέσουμε τα ελάχιστα πρότυπα. Φυσικά τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν τις ε, προδιαγραφές αυτές και να τις ε, εμπλουτίσουν. Χρειάζεται κατάλληλη συμβουλευτική εις βάθος λεπτομερής, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τεστ DNA και τα τεστ πρόγνωσης. Στην νέα διατύπωση υπάρχει μία διαφορά. Στα τεστ, για παράδειγμα, τα οποία απλά επιβεβαιώνουν μία ήδη ε, υπάρχουσα διάγνωση. Μόνο όταν ε, διαπιστώνεται μία γενετική ασθένεια, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση. Η διάγνωση όμως δεν πρέπει να δίδεται χωρίς σε μία διεξοδική συμβουλευτική. Διότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτά που θα λέμε στους ασθενείς. Ένας 18χρονος, για παράδειγμα, που ενημερώνονται ότι στο μέλλον θα νοσήσει από μια βαριά ασθένεια. Είναι κάτι που επιφέρει συνέπειες. Τώρα, πρέπει να έχουμε όσο βάση μας την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσον αφορά τις επιποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους οργανισμούς πιστοποίησης. Και όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους ε, συναδέλφους, να πω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η Ρεβέκα αναφέρθηκε στις εσωτερικές δοκιμές και πιστεύω πως πραγματικά μας έδωσε μια πολύ καλή βάση για να καταλήξουμε σε έναν οριστικό συμβιβασμό. Δεν θέλουμε. Τα τεστ που διατίθενται στο εμπόριο να χρησιμοποιούνται από τα νοσοκομεία χωρίς πρώτερη έγκριση. Όταν όμως δεν υπάρχουν κάποια τέτοια τεστ διαθέσιμα στο εμπόριο, για παράδειγμα για βαριές μεταδοτικές ασθένειες. Εδώ πρέπει να προβλέπετε κάποια εξαίρεση και πιστεύω ότι το κείμενο της Ρεβέκα Τέιλιορ πραγματικά αντανακλά αυτά που θέλουμε να προσθέσουμε. Αναφέρεται δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μεν λεπτομέρειες αλλά όχι γραφειοκρατία. Επίσης, μια πρόταση, υπάρχει μια πρόταση η οποία ορίζει τα νέα προϊόντα, διαγνωστικά προϊόντα και τα ταξινομεί στην κατηγορία D. Να πω ότι δεν ξέρω και τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μέχρι τώρα δεν είμαι σίγουρος για το αν αυτό μας καλύπτει όσον αφορά την ασφάλεια για τα πρώτα υψηλού κινδύνου. Τώρα, όσον αφορά τους συνοδούς διάγνωσης, τους, ε, τα τεστ δηλαδή που παρέχουν πληροφορίες για το αν μια συγκεκριμένη θεραπεία θα έχει αποτέλεσμα σε έναν συγκεκριμένο ασθενή. Εδώ πρέπει να συμπεριληφθεί και η άποψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Το ζήτημα είναι πώς. Ίσως πρέπει να συμπεριληφθεί στον ορισμό των κοινών ελάχιστων προτύπων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα ολοκληρώνω η διαφάνεια και το ζήτημα της Επιτροπής Διοντολογίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, κλινικές ε, δοκιμές και τις μελέτες κλινικών επιδόσεων. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει και στην ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Και φυσικά πρέπει να αξιολογήσουμε όντως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ε, της απογευματινής και να το συμπεριλάβουμε στις τροποποιήσεις μας. Φυσικά και χρειάζεται διαφάνεια, πρέπει όλοι να είμαστε ενημεροί για το τι συμβαίνει. Τώρα όσον αφορά την απόλυτη διαφάνεια, το θέμα εδώ, το ζητούμενο είναι πού βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στην απόλυτη διαφάνεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσπαθήσαμε να βρούμε συμβιβαστική λύση, πιστεύω πως έχουμε μια καλή αφετηρία. Και τώρα όσον αφορά την ε, Επιτροπή Δεοντολογίας, πρότεινα κάτι διαφορετικό από, ότι, από αυτό που συζητήσαμε. Χρειάζεται φυσικά να συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να βρεθεί ένα σε λιγότερο γραφειοκρατικός τρόπος παράκαμψης του προβλήματος. Η Επιτροπή Διοντολογίας θεωρώ πως είναι προβληματικό να ασχολείται με, την, με μια έκθεση, μια μελέτη τέτοιου είδους. Πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση αντιμετώπισης. Αλλά όπως είπα θα δούμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σήμερα το απόγευμα και θα δούμε πώς θα συζητήσουμε. Χρειάζεται φυσικά αξιολόγηση αυτής της Επιτροπής Δεοντολογίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρώτα υψηλού κινδύνου για τους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ Πετρελίζε. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω ορισμένους ε, καλεσμένους από τη Βόρεια Ιρνανία Βεσφαλία, του SPD, των Σοσιαλιστών. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Συνεχίζουμε τώρα την συζήτηση. Ο λόγος στους σκιώδεις εισηγητές. Dagmar Ευχαριστώ πολύ, Μαθίε. Είναι πολύ καλή η έκθεση του κυρίου Λίζε και η ελπίδα μου είναι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα επί τη βάση αυτής της έκθεσης. Έχω βέβαια καταθέσει πολλές τροπολογίες. Και είναι και τροπολογίες που έχω καταθέσει και στη δική μου έκθεση ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορία D των προϊόντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro. Βέβαια είναι καλύτερη κατάσταση από ό,τι στη δική μου έκθεση. Νομίζω ότι η ταξινόμηση γίνεται πολύ καλά στην πρόταση της Κομισιόν και συμφωνώ με τον Πέτερ Λίζε για το θέμα της θέσης σε ισχύ και του χρονοδιαγράμματος ότι είναι απαραίτητο να το επανεξετάσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Λίζα έχει καταθέσει και μερικές περαιτέρω τροπολογίες που αφορούν το θέμα της κατηγορίας D και, ορισμένα, και με τα ορισμένα προϊόντα της κατηγορίας C. Αυτό αντανακλά αυτό που είπαμε και στο παρελθόν, ότι ακόμα και η οι <clears throat> διαδικασία δοκιμασίας από τους ίδιους τους παρασκευαστές πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρουμε αν ένα τέτοιο τεστ μπορεί πάντα να καταδείξει αν μπορεί να υπάρξει ένας κίνδυνος μόλυνσης ή αν ε, τελικά το, η δοκιμασία αυτή θα λειτουργήσει πολύ διαφορετικά στην πράξη από ό,τι στο εργαστήριο. κύριος Λίζε ε, τονίζει τη σημασία των διαδικασιών και ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται μόνο κατόπιν συνταγηγόγραφησης. αλλά για μένα είναι σημαντικό ότι τα συνοδευτικά, οι συνοδευτικές δοκιμασίες θα πρέπει και αυτές να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο. Έχουμε ορισμένες τροπολογίες που προβλέπουν μια διαδικασία παροχής συμβουλών και κατά τα λοιπά νομίζω ότι είναι πολύ καλή η κατεύθυνση της έκθεσης. Μπορούμε να σταθούμε ίσως πιο προσεκτικά στην τροπολογία 5 και 7. Εκεί αναφέρω ότι το σημαντικό είναι για μένα αυτό το οποίο έχει καταδειχθεί από την πραγματικότητα ότι πρέπει να υπάρξει μια πληροφορημένη έγκριση κατά κάποιο τρόπο να γίνεται με πλήρη γνώση και κατανόηση του ασθενούς η δοκιμασία, η κάθε και ελπίζω ότι εδώ η έκθεση του κυρίου Λίζε η οποία αφορά μια πολύ ειδική ε, κατηγορία ιατροτεχνικών προϊόντων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα θα πρέπει εδώ να βρούμε μια βασική λύση και ελπίζω θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία για τα θέματα αυτά των κλινικών δοκιμασιών in vitro. Η Ρεμπέκα Τάιλερ έχει τώρα το λόγο σκιώδη συγγήτρια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ, εν συντομία, θα εκθέσω τις προθέσεις μου μέσω των τροπολογιών που κατέθεσα για την πρόταση για τα, σε, την in vitro διάγνωση. Ε, σε σχέση με τη διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό η νομοθεσία να είναι διαφανής και να εστιάζεται στον ασθενή και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων έτσι ώστε οι επαγγελματίες αλλά και το ευρύ κοινό να μπορεί να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Κατέθεσα κάποιες τροπολογίες εδώ για τη διευκρίνηση ε, των ε, κλινικών ε, μελετών και της απόδοσης που θα είναι διαθέσιμα μέσω της βάσης δεδομένων, πράγμα που δεν ήταν απόλυτα σαφές από την πρόταση της Κομισιόν, σε σχέση ε, με την ασφάλεια των ε, ε, ασθενών. Ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση της, του κόσμου συνδε, για να υπάρχουν στοιχεία για την επαγρύπνηση, φαρμακοεπαγρύπνηση και για να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού των προϊόντων σύντομα, πιο γρήγορα. Σε σχέση με τη διακυβέρνηση προσπάθησα να αναφερθώ στο σύστημα των κοινοποιημένων οργανισμών που χρειάζονται κάποιες αλλαγές για να ε, ε, υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα και πιο αυστηρή νομοθεσία. Δύο από αυτές προτείνουν μεγαλύτερη εξουσία αφορά την αναστολή κοινοποιημένων οργανισμών που δεν ανταποκρίνονται στα μήνυμα προδιαγραφές και επίσης να δημιουργηθεί μια ομάδα συντονισμού ώστε να είναι υποχρεωτική η έρευνα ε, για συγκεκριμένους κοινοποιημένου οργανισμού, από τη στιγμή που η ομάδα περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει ε, ζητήσει κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκού επίπεδου έλεγχο των κοινοποιημένων οργανισμών, συστήματα για να αυξηθεί η ανιχνευσιμότητα, αλλαγές που ξεπερνούν το καθεστώς αυτός και αυτό που ισχύει σήμερα και είναι ευπρόσδεκτες αλλαγές. Σε σχέση με τις τροπολογίες τώρα που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, να πω ότι υπάρχουν διάφορες τροπολογίες της Dagmar Rothbard που ελπίζω πω θα γίνουν δεκτέ από την Επιτροπή συμπεριλαμβανομένων των ε, διατάξεων περί ε, των νομοθετημάτων μάλλον περί διαφάνειας των κοινοποιημένων οργανισμών ώστε οι κατασκευαστές να πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή όταν ζητούν ε, μάλλον όταν ζητούν άδεια από κάποιο κοινοποιημένο οργανισμό σε άλλο κράτος μέλος. Δεν είμαι βέβαιος τώρα αυτό πώς θα το, εξασφα... Βέβαια πώς θα το εξασφαλίσουμε. Ο εισηγητής το ανέφερε. Ε, το γνωρίζει και τη δική μου προσέγγιση και την έχει στηρίξει πολύ, καθώς και οι υπόλοιποι σκιώδεις εισηγητές. Ε, νομίζω πως η διατύπωση που κατέθεσα στην τροπολογία 138, 141 και 142, μαζί με τους συναδέλφους ε, ε, Μακάβαν και Γιανακουδάκης, δίνει μια μέση λύση που είναι μια καλή επιλογή για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μαργαρέτα Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω και εγώ ορισμένα σχόλια. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πετρελίζε για την εξαιρετική <laughs> συνεργασία που είχαμε, καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τις εξαιρετικές προτάσεις τους. Καταρχάς, όσον αφορά τα τεστ αυτοδιάγνωσης. Με ανησυχεί λίγο το γεγονός ότι κανείς άλλος δεν τόνισε αυτόν τον τομέα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, αν έχει ένα λάθος αποτέλεσμα σε τεστ HIV, έχει πολύ σοβαρές συνέπειες, όπως επίσης και τα πιεσόμετρα. Εάν υπάρχουν λάθος αποτελέσματα τότε ενδέχονται να υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπλοκές σε μελλοντικές θεραπείες με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Τα τεστ αυτά δεν είναι πάντα αξιόπιστα και υπάρχουν ορισμένα βέβαια τεστ τα οποία φαίνονται απλά, για παράδειγμα μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα, όμως πραγματικά τα λάθος αποτελέσματα μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε υπάρχει η δική μου τροπολογία όσον αφορά την καλή συμβουλευτική για τα τεστ αυτά. Και τώρα όσον αφορά τις εσωτερικές δοκιμές, να πω ότι με βρίσκουν πολύ ικανοποιημένοι οι τροπολογίες που έχουν προταθεί για τις εξαιρέσεις, όμως να πω ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται εις βάρος του καλού των ασθενών. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα παραθυράκι στην νομοθεσία το οποίο να επιτρέπει την κυκλοφορία προϊόντων υψηλού κινδύνου στην αγορά. Όσον αφορά την έγκριση για κυκλοφορία στην αγορά. Δεν συμφωνούμε όλοι για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, όμως σίγουρα συμφωνούμε με το ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στο πώς πρέπει να διατίθενται στην αγορά τα προϊόντα υψηλού κινδύνου οι ασθενείς δεν πρέπει να είναι εκείνοι που θα πληρώσουν το τίμημα, παρά μόνο οι κατασκευαστές. Και όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, που είναι κάτι που θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα, ο κύριος Λίζε ήδη αναφέρθηκε σε αυτό και η Ντάγμα έχει καταθέσει τη δική της τροπολογία, η οποία πιστεύω πως πράγματι βελτιώνει την ασφάλεια των πολιτών και πιστεύω πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποχωρήσουμε στα εμπορικά συμφέροντα. Και σε σένα πηγαίνει αυτό, Πίτερ. Θέλω να με ακούσεις, σε παρακαλώ. Χθε η φαρμακευτική βιομηχανία στη Δανία απευθύνθηκε σε όλους εμάς και μας είπε ότι πραγματικά όλες αυτές οι απαιτήσει για περισσότερη διαφάνεια είναι ανοησίες. Είναι ψέμα αυτό. Είναι ξεδιάτροπο ψέμα και όταν αναφέρονται εκείνοι σε διαφάνεια, δεν είναι, δεν είναι διαφανής η διαδικασία, όχι, αναφέρονται σε ιδίους πόρους. Πραγματικά Παίζονται πολλά εδώ. Και το λέω στα αγγλικά, διότι τα γερμανικά μου δεν είναι καλά, αλλά να σου πω ότι όταν του ζητήσαμε να μας δώσουν παραδείγματα, τα παραδείγματα νομίμων συμφερόντων, τα οποία θα είναι τόσο σημαντικά ώστε να παρακαμφθεί η υγεία των ασθενών, δεν μπόρεσαν να μας δώσουν ούτε ένα επιχείρημα. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα και υπάρχουν και συνάδελφοι εδώ οι οποίοι τα προασπίζονται. Αλλά πραγματικά, όταν τους ζητούμε να μας δώσουν αυτά τα επιχειρήματα, δεν μας απάντησαν τίποτα. Να το λάβετε λοιπόν αυτό υπόψη διότι πραγματικά η φαρμακευτική βιομηχανία είναι τόσο σίγουρη ότι σήμερα το απόγευμα τα συμφέροντά τους θα υπερτερήσουν έναντι των, του συμφέροντος των ασθενών, που πραγματικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και Ντάκμαρ, σε ευχαριστώ πολύ που στη δική σου έκθεση ήσουν σαφέστατη. Ελπίζω να είμαστε ενωμένοι σήμερα το απόγευμα, έτσι ώστε να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για τα ξεκάθαρα λόγια σου, Μαργαρέτα. Μίλαν Κάρπνο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αν δούμε το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και τη σχέση με την οδηγία για τα ιατροτεχνικά Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και οι προτάσεις για γλωσσική απλοποίηση στα κείμενα και την διοικητική, διοικητική απλοποίηση. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα. Τώρα το να μπορούμε να εξαιρέσουμε από τις ε, συσκευές in vitro αυτές που δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη λειτουργία του ιατροτεχνικού προϊόντος και η, η διαδικασία αυτή Και είναι απαραίτητο λοιπόν να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα ρυθμίσουμε την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση των ε, ιατροτεχνικών συσκευών και όχι να τις, ε, τις περιλάβουμε στο τωρινό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Η Άλτα Σούζα για την ΚΟΕ. Eh, Σας ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον Πίτερ Λίζε ε, για την έκθεση που έκανε. Υπάρχουν σημεία που συμφωνώ και που διαφωνώ, όμως ο μέθοδος εργασίας που ακολούθησε ήταν ε, πολύ καλή γιατί επέτρεψε να υπάρξει μια παρασκευαστική φάση ε, για την έκθεσή του. Συζήτησε με τους κοιόδης για να μπορέσει ήδη να συμπεριλάβει κάποια σημεία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με διάφορα σημεία που ενέφερε και που μάλιστα εκείνος εισήγαγε στην έκθεση για παράδειγμα οι πτυχές που αφορούν τις γενετικές δοκιμές και το γεγονός ότι οι κλινικές δοκιμές που σχετίζονται με την in vitro διάγνωση υποχρεώνουν στην θετική γνώμη της ε, Επιτροπής ε, Ηθικής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το ψηφίσουμε απόψε σε ένα άλλο θέμα που είναι το, ο φάκελος των κλινικών δοκιμών. Πιστεύω επίσης ε, πως γεγονός ότι αναφέρονται τα, οι συνοδοί ε, των τεστ στα εργαστήρια είναι πολύ θετικό. Φυσικά, μεριμνώντας ώστε να εγγυηθούμε να μην σημαίνει αυτό καμία εμπορική συναλλαγή, ότι δηλαδή με αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο πολύ συχνά και στο γενετικό ε, πλαίσιο για την ε, έρευνα σε σπάνιες ασθένειες <coughs> γίνονται δοκιμές ε, ε, και μετά δεν υπάρχει εμπορευματοποίηση των ε, προϊόντων ή των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες τις οποίες εισήγαγε τώρα η ομάδα μου. Εκεί περιλαμβάνεται η ιδέα να αποσαφινιστούν κάποιοι ορισμοί, ιδιαίτερα οι ορισμοί που αφορούν τις ιδιαιτερότητες και την πρόσβαση, καθώς και την κλινική εγκυρότητα και την ε, κλινική αξία που δεν, νομίζω πως δεν ε, διευκρινίζονταν αρκετά ξεκάθαρα στην αρχική πρόταση. Επίσης, κατά την άποψή μας, η τάξη γάμα των προϊόντων αυτών θα πρέπει να θεωρείται μία τάξη υψηλού κινδύνου και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι είμαστε υπέρ αδειοδότησης πριν να τεθεί στην εμπορία. Το ίδιο όπως και για τους, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Δεν βλέπω να υπάρχει λόγος δηλαδή να υπάρχει εδώ διαφορά. Θα πρέπει να γίνει παράλληλη εργασία, γιατί πιστεύω πως ε, και τα δύο θέματα είναι σχετικά. Φυσικά είναι διαφορετικό να τοποθετεί κανείς ένα φύτευμα εντός του σώματος από το να κάνει ε, μια διάγνωση, αλλά και να έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την υγεία ή για την εξέλιξη της υγείας των ατόμων. Γι' αυτό οι εγγυήσεις που θα πρέπει να καλύπτουν αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να είναι όσο γίνεται ψηλότερο επίπεδο. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Πιστεύω πως θα έχουμε βέβαια μπροστά μας πολλή δουλειά ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να είναι συμβατέ οι δύο οδηγίε που εξετάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ δύο ακόμα ομιλητές, Ιάννε Ρόσπαχ και η κυρία Μαγκίνε. Υπάρχει κάποιο άλλο ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο και δεν τον είδα. Όχι. Κλείνω το κατάλογο, Ιάννε Ρόσπαχ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μείνουμε ιδιαίτερα τεχνική στα θέματα αυτά, Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λίζε για την τόσο καλή έκθεσή του. Είναι εξίσου εξαίρετη η έκθεσή του με την έκθεση της Ντάγμα ε, και συμφωνώ και με την κυρία Άουκεν για την αυτοδιάγνωση, τα αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες. Δεν πρέπει να κάνουμε διαγνώση για το DNA ή για άλλα θέματα στον εαυτό μας όταν δεν είμαστε εμείς ε, εμπειρογνώμονες. Είναι επίσης πολύ εύκολο να πάρει κανείς από το ίντερνετ αμφίβολης αξίας διαγνωστικά προϊόντα από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Εγώ πρότεινα την τροπολογία 144. Έχω ένα πρόβλημα με το τμήμα 4 της ε, τροπολογίας αυτής που κατέθεσα μαζί με άλλους. Δεν ξέρω αν δημιουργούμε εδώ πέρα ένα παραθυράκι και αναφέρομαι για τις, για τις νεαρές ε, μέλουσες μητέρες που είναι 14, 15, 16 χρονών. Εάν πρόκειται για γενετική ε, δοκιμασία πρέπει να αποφασίσουν αυτές ή οι γονείς τους. Είναι αυτό μια, ένα παραθυράκι το οποίο έχουμε ε, παραγνωρίσει ή είναι υπερβολικό αυτό που σας λέω. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ίδια τροπολογία, την 144, και να στηρίξω την πρόθεσή της, διότι Πιστεύω πως οι γενετικές δοκιμές και οι δυνατότητες να δώσουν αποτελέσματα στον κόσμο πρέπει να ελέγχονται πολύ προσεκτικά. Το θέμα δηλαδή της ενημέρωσης για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, γενετική, συμβουλευτική και το θέμα περί ανηλίκων. Η κυρία Ρόσμπακ έθιξε ένα ιδιαίτερο σημείο που ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά. Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε παραθυράκι. Πάντως είναι πρόκληση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα όταν πρόκειται για ανηλίκους. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά τις γενετικές δοκιμές. Ιδιαίτερα αν αυτό καλύπτει προβλήματα που δεν έχουν λύσει. Η πρόκληση είναι να αντιμετωπίσουμε τη δυνατότητα της τεχνολογίας να προβλέψει ε, προβλήματα υγείας. Και γι' αυτό και πιστεύω πως αυτή η τροπολογία 144 είναι καλά συνταγμένη για να αντιμετωπίσει το θέμα παρά το προσχόλιο της κυρίας Ρόσμπακ όσον αφορά τις ε, ανήλικες μητέρες. Το στηρίζω. Ε, πιστεύω πως είναι σημαντικό και η τελευταία παράγραφος της τροπολογίας είναι ε, επίσης σημαντική γιατί προβλέπουμε για τα μέλη, κράτη-μέλη που μπορούν να πάνε πιο μακριά από αυτή τη διάταξη και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω τώρα το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους Ευρωβουλευτές για την εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση Πραγματικά μαθαίνουμε τους λόγους πίσω από τις τροπολογίες και αυτό θα βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει αυτό το θέμα. Όσον αφορά την προέγκριση για την κυκλοφορία στην αγορά, έχουμε ήδη αναφέρει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα πλαίσια της προηγούμενης έκθεσης. Δεν θα επαναληφθώ λοιπόν εδώ. Καταλαβαίνουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι το θέμα των in vitro διαγνωστικών τεστ και τις πληροφορίες ε, σχετικά με αυτά. Τα τεστ αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς πληροφορίες έτσι ώστε, ο ασθενή να είναι πλήρως ενήμερος. Αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια, έχει να κάνει με ζητήματα δεοντολογίας, διότι πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να διασφαλίζεται μόνο η ασφάλεια του προϊόντος, αλλά και το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Πραγματικά λοιπόν είμαστε στη διάθεσή σας για βοήθεια σε οτιδήποτε τεχνικό και άλλα θέματα όσον αφορά τη συνταγογράφηση. Αυτό είναι κάπως ε, περίπλοκο νομικά η αφετηρία αυτών των ε, τροπολογιών, δηλαδή των απαιτείται συνταγή γιατρού για τη χρήση ορισμένων αυτών προϊόντων, είναι κάτι το περίπλοκο διότι υπάρχει αρχή της επικουρικότητας, υπάρχουν τα προνόμια που έχουν τα κράτη-μέλη σε αυτόν τον τομέα. Το να βρεθεί λύση λοιπόν είναι κάτι περίπλοκο. Βλέπουμε το όφελος ορισμένων προτάσεων από τους ευρωβουλευτές. Μερικά παραδείγματα θα σας δώσω ενδεικτικά. Πώς δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε για παράδειγμα την ε, πρόσβαση σε πληροφορίες σε κλινικές δοκιμές. Φυσικά είναι αναγκαία η ισορροπία εδώ. Υπάρχουν ωφέλη σε πολλές προτάσεις, η ανάμειξη των ενδιαφερομένων, των φορέων, η σύγκριση των ε, τελών, η συμβατότητα των ε, προϊόντων αυτών με άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορου ενδιαφερόμενους. Η πρόταση αυτή έχει πραγματικά πολλά αξιόλογα στοιχεία και όσον αφορά τι επιτροπέ δεοντολογίας να σα υπενθυμίσω ότι πρέπει να εναρμονιστούμε και με αυτά που κάνουμε στην πρόταση για τι κλινικέ δοκιμέ. Σε γενικέ γραμμέ πιστεύω να βρήκατε χρήσιμε όλε αυτέ τι προτάσει και είμαστε στη διάθεσή σα για περαιτέρω συνεργασία πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συγητής έχει τέλος το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις, ε, τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Θα ήθελα να κάνω σαφές και πάλι ποια είναι η οδηγός γραμμή της πρότασής μου. Η Dagmar Rothbeder τόνισε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας αν υπάρχει κάποια αμφιβολία για κίνδυνο μόλυνσης, αυτό είναι κάτι διαφορετικό με το να έχει κανείς μια λανθασμένη διάγνωση η οποία μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του. Εμείς τονίζουμε τη σημασία να υπάρχουν πρότυπα για τα in vitro test, ακόμα και αυτά τα οποία δεν μπορούν να έχουν τόσο σημαντικές συνέπειες λόγω μόλυνσης για την ανθρώπινη υγεία. Όλα αυτά πρέπει να τύχουν αυστηρής, αυστηρού ελέγχου <clears throat> και φυσικά ο ιατρός πρέπει να χρησιμοποιήσει και άλλες ε, μέρημνες στην ε, διάγνωση αλλά πρέπει όταν υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν σοβαρές συνέπειες να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που αναφέρθηκαν στην κατηγορία 4, στην κατηγορία D. και ότι εκεί πρέπει να υπάρχει μια συνολική κοινή διαδικασία. Τώρα η Κομισιόν φαίνεται να έχει κάποιες αμφιβολίες γιατί υπάρχει και πρόβλημα με την επικουρικότητα. Όλα αυτά ίσως πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση. Ξέρω ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν κάποια προγράμματα για να αντιμετωπίσουν ομάδες κινδύνου του HIV, παραδείγματος χάρη, ή άλλες περιπτώσεις για να υποβάλλονται σε δοκιμασίες και αυτό είναι μια εξαίρεση η οποία μπορεί να ισχύσει επί τη βάση αυτής της επικουρικότητας. Και, αλλά, κατά τα άλλα, οι τροπολογίες 111 και άλλες που αφορούν αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν με το Συμβούλιο. Για τη διαφάνεια. Μαργαρέτε, έχεις δίκιο αλλά το ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους ε, ε παραγωγούς βασμάτων με τη διαφάνεια. Όσοι έχουν γνωρίσει την ιστορία του Βιόξ, αυτό είχε παρουσιαστεί ως ένα αναλγητικό χωρίς παρενέργειες. Ενώ σήμερα ξέρουμε ότι η διαδικασία κλινικών μελετών, μελετών δεν ήταν διαφάνεια και αν δεν ήταν διαφανής και αν ήταν διαφανής τότε μάλλον δεν θα είχε ποτέ εγκριθεί αυτό. Υπάρχουν διαδικασίες λοιπόν οι οποίες δεν είναι επαρκείς και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στους τομείς αυτούς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δίδονται τα στοιχεία για τις ε, κλινικές αυτές μελέτες, για τα προϊόντα in vitro και θα πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητα τα αποτελέσματα αυτά. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες θα πρέπει οι εκθέσει να δημοσιεύονται. Εγώ έχω από την άλλη πλευρά τώρα ένα πρόβλημα με την εμπιστευτικότητα των στοιχείων για τους ασθενείς και με, ε, με, το απόρριτο των επιχειρήσεων πολλές φορές. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αντιμετωπίσει το γεγονός ότι πολλές φορές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πάρει στοιχεία εμπιστευτικά μικρών, μικρό και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο να λάβουμε υπόψη μας. Και εγώ φυσικά υποστηρίζω μεγαλύτερη διαφάνεια από ό,τι πριν, αλλά βέβαια η απόλυτη διαφάνεια θα προσκρούσει σε ορισμένα όρια για την τροπολογία 144. Ε, εγώ υποστηρίζω για την υποστήριξη που έλαβε. Η περίπτωση που ανέφερε η Άννα Ρόσπαχ για τις ε, νεαρές μέλουσες μητέρες, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί και στις εθνικές νομοθεσίες. Είναι φανερό ότι όταν πρόκειται για ένα ανήλικο άτομο, θα πρέπει να λάβει μεν την απόφαση, αλλά θα πρέπει να τύχει και της απαραίτητης παροχής συμβουλών. Αλλά αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπόκειται στι εθνικές νομοθεσίες που έχουν διαφορετικές <clears throat> ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την πρακτική που ακολουθούν αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το άτομο το οποίο πρέπει να πάρει την απόφαση είτε είναι οι ανήλικοι ή οι γονείς της θα πρέπει να τύχουν τις κατάλληλες παροχή συμβουλών. Επίσης, το σημείο 7 εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε όχι μια πλήρη εναρμόνιση, αλλά ελάχιστα κοινά πρότυπα, αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει δεκτό αυτό από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και η τροπολογία της κυρίας Βάις για ένα θέμα το οποίο το βλέπω πολύ θετικά αλλά και πάλι πιστεύω ότι ίσως θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό το θέμα στα κράτη-μέλη και αυτό το κάνω σαφές με μια αιτιολογική σκέψη. Τέλος, για τη διαδικασία δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε χωρίς λόγο την διαδικασία. Φυσικά είναι ένα ευαίσθητο θέμα και έχουμε συμφωνήσει μεταξύ των εισηγητών ότι μετά από την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε το ταχύτερο δυνατό σε μια, μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια αλλά χωρίς να κάνουμε τελική ψηφοφορία, χωρίς πρωτού τελειώσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Συνήθως εμείς κάνουμε μια διαδικασία μόνο μέχρι την πρώτη ανάγνωση ή φτάνουμε ως το τέλος, αλλά νομίζω ότι αυτή η διαδικασία του να αφήσουμε κατά μέρο την τελική ψηφοφορία μετά την Ολομέλεια, αυτό επιτρέπει να υπάρξουν διορθώσει. έχει αποδείξει την αξία τη αυτή η διαδικασία σε άλλε επιτροπέ. και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με τη Λιθουανική Προεδρία να καταλήξουμε σε ένα οριστικό ε, αποτέλεσμα. Θα μας δώσει περισσότερο χρόνο για και περιθώριο για διαπραγμάτευση χωρίς να καθυστερήσει ιδιαίτερα τα πράγματα αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ Πίτερ Λίζε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την συζήτηση. Μας μένει η ψηφοφορία. 10 Ιουλίου ψηφοφορία. Ενδεικτικά τον Σεπτέμβριο του 2013 θα πάει η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια. Με αυτό λοιπόν προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 7. Γενική έκθεση για τον κανονισμό REACH και επανεξέταση ορισμένων στοιχείων του. Περιμένουμε να έρθει ο κύριος Ντάνσερτ, η Κομισιόν είναι ήδη εδώ. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Πρέπει να δω τα ταμπελάκια για να δω πώς σας λένε. Βίλμοτ σας λένε, έχουμε και μία συνάδελφο. Καλώς ορίσατε λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Ντάνσετ και λοιποί. So, ich begrüße auch ganz herzlich. Καλώς ορίζω λοιπόν τον Κέρ Τάνσερτ, εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε. Προβλέπετε στο χρονοδιάγραμμα καταρχάς μία παρουσίαση της γενικής έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα συζήτηση και στο τέλος η παρουσίαση του κυρίου Τάνσερτ την οποία θα συζητήσουμε μετά θα ελάβουν το λόγο οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές. Καλώς ορίσατε λοιπόν, βλέπω γνώριμες φυσιογνωμίες εδώ στην Επιτροπή. Και Λαμπερότσο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρωτού πω σε λεπτομέρειες, να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημολογήσει μια πρόταση, έχει παρουσιάσει στον Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη για το 7ο πρόγραμμα δράσης το οποίο θα οδηγήσει σε ένα μη τοξικό περιβάλλον. Και η REACH είναι ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο του προγράμματος αυτός και τονίζεται λοιπόν η σημασία του και η ανάγκη για περαιτέρω δράσεις όσον αφορά τις μίξεις χημικών και τις επιπτώσεις τους αυτές στα προϊόντα και στο περιβάλλον. Συνολικά, ο σκοπό του ΡΙΤΣ είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασία στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο της ε, στρατηγική μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και η ευκαιρία λοιπόν που έχουμε να το συζητήσουμε αυτό με την Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντική. Το συμπέρασμά μας από, την αυτή, από αυτή την αξιολόγηση είναι ότι το REACH έχει αποτελέσματα. Οι στόχοι οι οποίοι θέσαμε βρίσκονται σε καλό δρόμο. Δεν έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε όλους τους στόχους, αλλά τουλάχιστον επιτύχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Και σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι πραγματικά έχει αποτελέσματα το REACH αυτό και το κύριο συμπέρασμα. Κοιτάξαμε λεπτομερώς το αν υπάρχουν κάποια κενά ή κάποιες αλληλοεπικαλύψεις στο νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τα χημικά προϊόντα. Δεν βρήκαμε σε γενικές γραμμές κάτι τέτοιο, δεν εντοπίσαμε κάτι τέτοιο. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες να έχουν μια ασφάλεια και μια προβλεψιμότητα την οποία θα δώσει αυτό λοιπόν το σταθερό πλαίσιο. Προτείνω λοιπόν να μην γίνουν ε, μεγάλες ε, και σημαντικές τροποποιήσεις στις κύριες διατάξεις. Είδαμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για βελτίωση και ίσως να σας παρουσιάσω ορισμένες από αυτές. Καταρχάς οι προθεσμίες καταχώρησης που ισχύουν από το 2010. Σε γενικέ γραμμέ πιστεύουμε ότι ήταν κάτι που είχε επιτυχία, δεδομένου του αριθμού των ε, αιτήσεων που μας υποβλήθηκαν. Σίγουρα χρειάζονται βελτιώσει στην ποιότητα των αφακέλων που κατατίθεται από την βιομηχανία και η ΕΚΑ έχει εντοπίσει ορισμένες ε, περιπτώσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται πλήρως με τον κανονισμό. να ληφθούν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα βήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εντοπισμό, τον ακριβή εντοπισμό των ουσιών, οι οποίες πρέπει να τυχαίνουν καλύτερης ανάλυσης, καθώς και των ενδιάμεσων ουσιών, Τις επόμενες ημέρες ε, λοιπόν θα κοιτάξουμε λεπτομερώς ε, τις νέες ε, προθεσμίες καταχώρησης, προβλέπονται προς το τέλος του μήνα. Και θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την ταυτοποίηση των ουσιών αυτών. Η δεύτερη, ο δεύτερος τομέας βελτίωσης είναι η έγκριση και η διαδικασία έγκρισης για τις χημικές ουσίες. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών με λιγότερο επικίνδυνες. Ήδη από τώρα έχουμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι γίνονται έγκαιρες δράσεις για την αντικατάσταση των ουσιών αυτών και έχουμε λάβει και αιτήματα για τη βελτίωσή τους από πάρα πολλούς. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι επιτελείται πρόοδος όσον αφορά αυτό. Υπάρχουν αρκετές ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο προς έγκριση και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τους υπόλοιπους ε, φορείς προς την ολοκλήρωση ενός οδικού χάρτη με στόχο το 2020. Επίσης ένας άλλος τομέας που επιδέχεται βελτιώσεις είναι το αν πραγματικά θα καταφέρουμε να σπάσουμε τους φραγμούς στην ενιαία αγορά. Ήταν ένας από τους στόχους του κανονισμού REACH και πιστεύω πως έχουμε ορισμένες ενδείξεις που δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη διστάζουν να λάβουν μέτρα, όμως έχει παρατηρηθεί πρόοδος. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη πρόοδος για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της, του κόστους, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ στενά και με την υπηρεσία και με τα κρατη έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, ατομικούς χρήστες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επιμερισμό του κόστους. Σκοπεύουμε να οργανώσουμε ένα εργαστήριο επίσης για την αναθεώρηση του REACH στις 27 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε πλήρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε για το πώς λειτουργούμε. Το κεντρικό σημείο αυτού του εργαστηρίου θα είναι η ποιότητα των εφακέλων καταχώρησης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι ατομικοί χρήστες. Ο συνάδελφός μου τώρα, ο κύριος Βίλμοτ, θα σας ε, αναφέρει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βίλμοτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας <clears throat> για την Επιτροπή, για την ευκαιρία να μιλήσω για την αναθεώρηση του ΡΙΣ και ζητώ συγγνώμη για τον ε, ε Γενικό μου Διευθυντή, ο οποίος χρειάστηκε να, να αντιπροσωπεύσει τον κύριο Ταγιάννη σε μια άλλη εκδήλωση Πιστεύουμε λοιπόν, όπως είπε και ο συναδελφός μου, ότι το REACH λειτουργεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά βοηθάει και την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Να πω τώρα σε λίγο περισσότερο βάθος για την ανάλυση μας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. <clears throat> Δείχνει η έρευνά μα ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι οι μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις είναι πιο τροτές από τα αποτελέσματα του ΡΙΤΣ από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις λόγω και της οικονομικής κρίσης είναι πιο δύσκολο να μάθουν για το ΡΙΤΣ και να ενσωματώσουν το κόστος το οποίο απαιτείται για τη συμμόρφωση με το ΡΙΤΣ. Είδαμε επίσης ότι πολλές εταιρείε δεν γνωρίζουν τα καθήκοντά τους και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν βάσει του ΡΙΤΣ. Επιπλέον, μετά από την έρευνα αυτή που έκανε η Κομισιόν και έδειξε ότι οι επιχειρήσεις μικρομεσαίου χαρακτήρα δείχνουν, θεωρούν το ρίτσο ότι είναι ένα από τα δέκα σημαντικότερα στοιχεία επιβάρυνσης της εργασίας τους. Έχουμε καταλήξει ορισμένες κατευθυντήρες γραμμές για να αντιμετωπίσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε διευρυμένα στοιχεία πληροφορία σε σχέση με το REACH, τι χρειάζεται να κάνουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του REACH. Ένα πρώτο βήμα σχετικά ήταν η περαιτέρω μείωση των τελών που πρέπει να καταβάλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Ευρωπαϊκό Φορέα Χημικών Ουσιών. Είναι πια μικρότερο αυτό το επίπεδο των τελών από ό,τι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και βέβαια υπάρχει και μια καταληκτική προθεσμία για καταγραφή μέχρι το τέλος του, της εβδομάδας αυτής. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα όμως τα οποία θέλουμε να κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα έγγραφα κατεύθυνση που δίνουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τα κάνουμε πιο φιλικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους δώσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα συμμόρφωσης και να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους για την ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμένες ουσίες και επίσης περισσότερες πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα και πώς <clears throat> να μα επικοινωνούν μαζί μας για το θέμα της χρήσης αυτών των χημικών. Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και τη διαδικασία έρευνας και καινοτομία και θα δημιουργήσουμε και μεγαλύτερη ε, συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης θα ήθελα να μιλήσω και για την δική μας για την υπηρεσία για τον φορέα χημικών ουσιών. Νομίζω ότι έπαιξε ένα κεντρικό και κέριο ρόλο η ΕΚΑ στην τεχνική και διοικητική διαχείριση του ΡΙΤΣ Ιδίω για την εξέταση των φακέλων, ο ρόλο τη ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οδήγησε σε βελτίωση τη ποιότητα των φακέλων που υπευλήθησαν για χημικέ ουσίε. Είμαι σίγουρο ότι ο φορέα αυτό θα συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση και θα ενισχύσει περαιτέρω τι δραστηριότητέ τη προ την κατεύθυνση τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στα κράτη-μέλη. Πέραν τη αναθεώρηση, θα ήθελα να πω για τον οδικό χάρτη για την, ε, τον εντοπισμό των ουσιών που έχουν ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρα. Το 2010 ο κύριος Σταγιάννη και ο κύριος Ποτόνσκι είπαν ότι πρέπει να επιταχυνθεί η καταγραφή αυτών των ουσιών. Ο στόχος ήταν να φτάσουμε τις 130 ουσίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια των κρατών μελών και της ΕΚΑ. Ο στόχος μας τώρα είναι όλες αυτές οι ουσίες να μπουν στον κατάλογο μέχρι το 2020. Για να το κάνουμε αυτό μαζί με τα κράτη-μέλη έχουμε καθορίσει ένα οδικό χάρτη για τις ουσίες αυτές, τις λεγόμενες SDH, τις οποίες αντιμετωπίζουμε τώρα. Είχαμε πολύ καλή ε, υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων και τώρα φυσικά πρέπει να υλοποιηθούν όλα αυτά. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δούμε να δούμε τις διάφορες ουσίες αυτές. Έχουμε καταρχήν τις ουσίες που είναι καρκινογενείς, ε, μεταλλαξιογενείς και καρκινογενείς. Επίσης ουσίες που είναι βιοσυσσωρεύσιμες και τις πάρα πολύ ε, επικίνδυνες ουσίες οι οποίες είναι ε, μη αποδομήσιμες κτλ. Μια δεύτερη ομάδα είναι οι ουσίες οι οποίες έχουν αντί, ισοδύναμο αποτέλεσμα όπως είναι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες κτλ. Όλες αυτές οι ουσίες, οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία είναι οι πιο σημαντικές από όλες. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε για τις ιδιότητές τους και για τις χρήσεις τους για να μπορέσουμε να καθορίσουμε την κατάλληλη αντιμετώπιση βάσει του ρίτσου, βάσει άλλων νομοθετημάτων. Το δικός χάρτης δημιουργεί και το σχέδιο δράσης για την Κομισιόν και την ΕΚΑ για να μπορέσουμε μέχρι το 2020 να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ουσίες. Το πρώτο βήμα θα είναι ένα εργαστήριο που θα διοργανώσουμε, που διοργανώσαμε το 2013 ήδη, όπου συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη για τις συγκεκριμένες δράσεις που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Υπάρχουν και άλλα εργαστήρια τα οποία προβλέπονται και θα αρχίσει και η πραγματική εργασία. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την ορμή που έχουμε ε, αποκομίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Κομισιόν. Και ερχόμαστε τώρα στους συντονιστές. Ο κύριος Ζέμπερ για το ΕΛΚ. Πρώτος. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις δηλώσεις τους Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει σε νομοθετικό επίπεδο να ε, εδραιώσουμε το σύστημα REACH, το οποίο είναι πρώτο πόρο σε παγκόσμιο επίπεδο και νομίζω ότι είναι σημαντικό που λέει η Κομισιόν ότι λειτουργεί. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες ε, ελλείψεις. Εγώ παίρνω συνέχεια παράπονα από περιβαλλοντικές οργανώσεις που δι... διαμαρτύρονται για την ποιότητα των διαδικασιών και αναφέρονται σε ένα αριθμό ουσιών που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του REACH. Και από τη μία πλευρά, όπως λένε οι βιομηχανικοί κύκλοι, ε, υπάρχει ιδιαίτερη, ιδιαίτερο φορτίο εργασίας το οποίο προέρχεται από την εφαρμογή του REACH. Βέβαια, όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αυτό αφορά ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Θα πρέπει εκεί να βελτιωθεί η διαδικασία καταγραφής. Και μέχρι το 2018 θα φτάσουμε ένα κόστος της τάξης των 2,5 ε, δισεκατομμυρίων είναι λοιπόν ε, το μεγαλύτερο εργαλείο το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ στα θέματα αυτά. Επίσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η διατήρηση της ε, ασφάλειας των ουσιών αυτών. Εδώ έχουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πλήρης εξέταση όλων αυτών των θεμάτων μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό κόστος και οι, τα παράπονα ναι έχουν οδηγήσει σε μείωση των τελών αλλά η πραγματική ανάγκη για να συμμορφωθεί κανείς με την ε, ε, νομοθεσία του ΡΙΤΣ εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε αυτό το σύστημα πιο φιλικτό φιλικό προς τους χρήστες χωρίς να υπάρξει μείωση των προτύπων, να διατηρήσουμε όμως τα υψηλά πρότυπα, αλλά να το κάνουμε πιο πρακτικά εφαρμόσιμο. Και φυσικά η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το σύστημα είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν εμπειρογνώμονες, έχουν άτομα τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν τις προδιαγραφές του του αλλά εμείς θα πρέπει με εργαστήρια και με άλλες ενέργειες να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση με την συμμετοχή των διαφόρων ενώσεων που εμπλέκουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά σε αυτές τις επιχειρήσεις. Παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για τον τομέα αυτό που είναι και η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. και επίσης θα πρέπει να διευρύνουμε το REACH και σε μια ευρύτερη ε, τάξη ουσιών. Υπάρχουν ε, και άλλες επικαλυπτόμενες ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά και έχουμε πάντα προβλήματα σύγκρουσης ε, προδιαγραφών με τις, τα νομοθετήματα που αφορούν τη, τα απορρίμματα και τα απόβλητα και γι' αυτό εδώ το REACH θα μπορούσε να αποτελέσει και μια γέφυρα και προς τα νομοθετήματα αυτά και επίσης θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ενίο χώρο για την υποβολή παραπόρων. Αυτό θα μπορούσε να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν στην αλυσίδα ε, προμήθειας ε, των ουσιών αυτών. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί η Κομισιόν να τα σκεφτεί περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζέμπερ. Κύριε Μακέιβεν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή για τις πληροφορίες. Είναι πολύ ευχαριστώ αυτό που άκουσα για το εργαστήριο, διότι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου περιβαλλοντικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και μου επισήμαναν ακριβώς αυτά που αναφέρατε κι εσείς και την ποιότητα μάλιστα των φακέλων, κάτι το οποίο ήταν πρόβλημα, καθώς και, τον, ε, και τις επιπτώσεις ε, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους ατομικούς ε, χρήστες. Είμαι σίγουρη ότι στο εργαστήριο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτές τις ανησυχίες. Υπάρχουν όμως και ορισμένες πιο λεπτομερείς, πιο λεπτομερείς ζητήματα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Στην δική μου εκλογική περιφέρεια είχα ορισμένες περιπτώσεις ε, λάθος καταχωρήσεων επιχειρήσεων, όχι όμως ασκεμένου λάθους. Αυτές οι επιχειρήσεις έτσι είχαν συμβουλευτεί να πράξουν. Υπήρχε λοιπόν μια γενικότερη σύγχυση σε αυτέ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν ήξεραν ακριβώ ε, τι να κάνουν. Όσον αφορά τώρα την ταυτοποίηση και τον έλεγχο για το εάν μια εταιρεία έχει εγγραφεί κανονικά. Υπάρχουν τέλη καταχώρηση. Καλώ. Μετά όμω υπάρχουν και πρόσθετα τέλη, διοικητικά τέλη έτσι όπω ε, ονομάζονται κατανοώ ότι αυτό το διοικητικό τέλος ισχύει από τον Φεβρουάριο. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που μια εταιρεία έχει κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ήδη από τον Ιανουάριο. Τι γίνεται με αυτό το διοικητικό τέλος. και με το πρόσθετο κόστος που αυτό το διοικητικό τέλος επιφέρει. Τι θα πληρωθεί πρώτο, τι όχι. Μία περίπτωση μάλιστα υπάρχει οπου μία εταιρεία αναγκάστηκε να πάρει δάνειο για να πληρώσει λοιπόν αυτήν την διαφορά του κόστου των ε, πρόσθετων τελών. Και φυσικά όταν παίρνει δάνειο πληρώνεις και τόκους αυτό το δάνειο στις δόσεις. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και στα πρόσθετα κόστη αλλά και στα πρόστιμα. Τώρα, η προθεσμία του 2018 πιστεύω ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει ολόνα και περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν αίτηση καταχώρησης, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πόσο οικονομικά εφικτό θα είναι αυτό και ελπίζω στο εργαστήριό σας να παρουσιάσετε κάποιον μηχανισμό στήριξης για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, τι γίνεται με τις δοκιμές σε ζώα. Κανείς δεν το ανέφερε αυτό ακόμα. Έχει το ρίτσο επιπτώσει στις δοκιμές σε ζώα. Πώς το υπολογίζετε. Επίσης, όσον αφορά την αντικατάσταση, αναφέρατε κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό. Κάποια στοιχεία που έχετε συλλέξει, αλλά πότε περιμένετε να συλλέξετε και ακόμα περισσότερα στοιχεία. Όταν αποσύρεται ένα προϊόν από την αγορά, τι γίνεται, υπάρχει κάποιο αντικαταστάτη του. Ευχαριστώ πολύ. Λίντα Μακέιβαν, Κρι Ντέιβι, εκ μέρου των Φιλελεύθερων, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μια από τι επιτυχίε του Ρίτς μπορεί να μετρηθεί από το γεγονός ότι πολλοί μας, και δεν είμαι ο μόνος, πολύ λίγοι παίρνουμε λογογραφία για το ΡΙΤΣ. Αν θυμηθεί κανείς ε, τι πίεση ασκήθηκε, πώς λόμπι υπήρχαν ε, τη φάση προετοιμασίας και κρίσης του ΡΙΤΣ, αυτό είναι εντυπωσιακό. Διάφορα θέματα βέβαια αναφέρθηκαν ήδη, τα μικρομεσαίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το, η περιπλοκότητα της ε, καταχώρησης. Δεν έχω καμιά ιδέα πώς οι τελικοί χρήστες μπορεί να συμφωμορφωθούν προς όλες αυτές τις ε, απαιτήσεις και να τονίσω ότι όντως η ΕΚΑ, λένε τα λόμπι, δεν κάνει αρκετά ώστε να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις ε, που έχουμε προβλέψει εμείς, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των εναλλακτικών στις δοκιμές σε ζώα. Επιπλέον υπήρξαν δύο ερωτήσεις, μία για να ακολουθήσω τα όσα είπε Λίντα. Με χαρά άκουσα ότι ο κατάλογος των υποψηφίων ουσιών αναπτύσσεται έτσι όπως μας είπατε. Δε βέβαια οι ΜΚΟ έρχονται και λένε μα μόνο τρεις περιορισμοί έχουν ε, εισήχθει». μα δεν είναι απαραίτητο να εισάγεται περιορισμός. Αν υπάρχει πρόταση πως, θα, ε, πως επίκειται περιορισμός τότε οι εταιρείε ε, λαμβάνουν τα μέτρα τους θα βρουν μια λειτουργούσα εναλλακτική εκ των προτέρων. Έτσι λειτουργεί το σύστημα και σωστά. το θέμα είναι αν όλα αυτά αρκούν για λόγω της, των ανησυχιών που προέκυψαν μέσω της ε, εισαγωγής της οδηγίας. Και έπειτα υπάρχει ε, το σεμινάριο που, που προβλέπεται, αλλά η καθημερινή επαφή με τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους αυτών για τη λειτουργία του ΡΙΤΣ, εδώ έχω κολλήσει λίγο. Όσον αφορά συζήτηση που θα μπορούσε, πιθανές ερωτήσεις μάλλον που θα έπρεπε να τεθούν, μα αυτές είναι ερωτήσεις που καθημερινά θα έπρεπε να ε, θέτουν οι εταιρείε ε, σε εσά, ε, σε σχέση με εσά, για το πώς θα λειτουργήσει πιο εύκολα το σύστημα για τις εταιρείε μας, ας πούμε, και εσείς με τη σειρά σας να απαντάτε για το πώς το REACH μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και πιο φθηνά. Μπορείτε να σχολιάσετε λοιπόν τι γίνεται, πόσο είστε βέβαιος ότι απαντάτε με τρόπους που να είναι ωφέλιμοι προς τις επιχειρήσεις όταν αυτές σας προσεγγίζουν και σας θέτουν τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ε, το χάσει. Μια έμπειρο γνώμων στην ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που ήρθατε στην ε, Επιτροπή μας σήμερα. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτό το χρονοδιάγραμμα για να έχουμε όλες τις σχετικές ουσίες ε, που για τις οποίες ανησυχούμε μέχρι το 2020 πιστεύω ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ αργό. Ε, η νομοθεσία επιτέλους οριστικοποιήθηκε το 2006 και μιλάμε 11 ε, χρόνια phasing in, ενώ τώρα από ό,τι φαίνεται σχεδιάζεται 14 χρόνια πριν όλες οι σχετικές ουσίες να έχουν μπει στον κατάλογο υποψηφίων ε, ουσιών ψηλού κινδύνου, υψηλής ανησυχίας. Και έπειτα έχω και δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα που συζητούσαμε αρκετές φορές, την ποιότητα των στοιχείων. Έχουμε ακούσει ότι είναι στοχευμένη η συμμόρφωση των ε, φακέλων και εταιρείε που δεν ε, έχουν ντοσιέ που να είναι σύμμορφα θα ενημερώνονται με μέσω επιστολής. Και έπειτα είπατε ότι ε, σε περίπτωση που οι εταιρείε δεν έχουν ετοιμάσει σύμμορφα ντοσιέ, θα αποσύρετε του αριθμού ε, καταχώρηση. Και θέλω να ξέρω αν έχει γίνει αυτό για κάποια εταιρεία ή όχι. Έπειτα, επίσης, ε, αποφασίσατε να δημοσιεύσετε αποφάσεις που έχετε υιοθετήσει σε σχέση με την μη συμμόρφωση των ντοσιέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά που ε, δημοσιεύεται διαγράφεται τα ονόματα των εταιριών έτσι ώστε τελικά δεν ασκείται δημόσια πίεση για αυτές τις εταιρείες για να βελτιωθούν. Έχετε σκεφτεί τη δημοσίευση των ονομάτων των εταιριών και τη χρήση της δυνατότητας ε, άσκησης πίεσης από το κοινό ως έναν τρόπο για να πετύχουμε την μεγαλύτερη συμμόρφωση στα στοιχεία. Τρίτη ερώτηση που συνδέεται με την ποιότητα των ε, στοιχείων. Μια πενταετής έκθεση ε, έδειξε ότι μόνο το 20% των καταγεγραμμένων φακέλων περιλαμβάνουν στοιχεία για την ε, καρκινογόνο χαρακτήρα, την τοξικότητα και και αν ε, το κατά πόσο η ουσία είναι VPVB ή VPVP. Αυτό ε, για το ντοσιέ, αλλά ποιο είναι το ποσοστό των ουσιών όπου ακόμα δεν έχετε πληροφορίες για το αν είναι CMR ή PBD ή VPVD. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον. Αυτά, αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται ε, στα ντοσιέ για φέτος. Γιατί είναι βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για την ταξινόμηση των ουσιών. Για να δούμε δηλαδή κατά πόσο είναι υψηλής ανησυχίας ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Άννα Ρόσπαχ στη συνέχεια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα από τον κύριο Βέλμοντ ότι γίνονται εργασίε για να κατανοήσουμε τώρα τι επιπτώσει του ΡΙΤΣ. Αλλά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνουν οι υπηρεσίε για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει συνοχή ανάμεσα στο REACH και στο ROS, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν για το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, ε, να επαναλάβω και εγώ την ερώτηση της Chris Davis για τις δοκιμές σε ζώα. Τι κάνει η Κομισιόν για να μειώσει τα ποσοστά δοκιμών σε ζώα στα πλαίσια του REACH. διότι ολοένα και περισσότερες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν ε, για τις δοκιμές ε, σε ζώα και θα ήθελα να ξέρω εάν χρησιμοποιούνται αυτές οι εναλλακτικέ λύσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις επίσης όπου ορισμένες ουσίες μπορούν να δοκιμαστούν χωρίς να χρησιμοποιηθούν ζώα. Όμως η νομοθεσία ακόμα ζητά δοκιμές σε ζώα. Και επίσης τι γίνεται σε περίπτωση δοκιμών σε ζώα που είναι ήδη νεκρά. Που έχουν σφαγιαστεί δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ολοκληρώσαμε τον κύκλο των ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε ερωτήσεις και στον κύριο Ντάνσετ. Και έπειτα θα ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Ντάνσετ. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έρθω στα ερωτήματα για τα ζώα και τις δοκιμασίες της ζώα. Έχουμε τριών ειδών θέματα εδώ. Πρώτα απ' όλα, το λεγόμενο data sharing ήταν μια ρήτρα στην νομοθεσία που είχε σαν στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Sharing. Και οι... και χερικά αυτές οι ρήτρε για, την... Ε, για το διαμοιρασμό των δεδομένων θα βοηθούσαν καλύτερα το να μειώσουμε την... Ε, τις δοκιμασίες σε ζώα. Και έτσι υπήρξε κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά. Ένα δεύτερο θέμα είναι σε ένα τομέα όπου δεν υπήρξε πρόοδος ή τουλάχιστον η πρόοδος που μπορούσαμε να αναμένουμε και να προσδοκούμε. <clears throat> Για επιχειρήσεις που υποβάλλουν φακέλους με στόχο να καταγράψουν τι γίνεται για την ευμάρεια των ζώων, αλλά δεν υπάρχει, που υποκτές δοκιμές, αλλά δεν υπάρχει επαρκής ποιότητα στοιχείων για να καταδείξει ότι γίνεται ασφαλής χρήση δοκιμασιών όταν δεν υπάρχουν άλλες <clears throat> επιστημονικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι η επιστημονική επιχειρηματολογία έχει εδρεωθεί επαρκώς και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει την πρόοδο που ελπίζαμε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν λοιπόν με την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας. Είναι ένα σημείο το οποίο τόνισα ότι θα λάβουμε υπόψη μας στο εργαστήριο που θα γίνει και σε άλλες ευκαιρίες. Ένα τρίτο σημείο είναι τι γίνεται για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των εναλλακτικών δοκιμασιών. Και επενδύουμε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ένα κονδύλιο 300 εκατομμύριων ευρώ, σε προγράμματα που θα υποστηρίξουν την έρευνα για αναλλακτικέ μεθόδους δοκιμασία. και επίσης και ένα εργαστήριο αναφοράς για τέτοιες μεθόδους εναλλακτικού χαρακτήρα. Υπήρξε μεγάλη πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί τέτοιες μέθοδοι και έχουν επικυρωθεί σε διεθνές επίπεδο ώστε να είναι αποδεκτές από τον ΩΣΑ και άλλους διεθνείς φορείς. Υπήρξε λοιπόν κάποια πρόοδος για να βρούμε <clears throat> εναλλακτικέ μεθόδους, αλλά ακόμα θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια από την ερευνητική κοινότητα και τα ερευνητικά προγράμματα. Αυτό το οποίο όμως μας ενδιαφέρει είναι να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες από τις επιχειρήσεις και στον τομέα αυτό δεν έχουμε προχωρήσει απόλυτα. Είναι λοιπόν ανάμεικτη η εικόνα σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για, τα, για τις δοκιμασίες σε ζώα. Ο κ. Ζέμπερ έθεσε το θέμα της συνεκτικότητας μεταξύ της ε, οδηγίας για το ρίσκο και της οδηγίας για την ανακύκλωση και επανάκτηση. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που έχουν ανησυχίες για τα θέματα αυτά. Έχουμε δώσει κάποιες κατευθυντές γραμμές για ορισμένες μορφές πλαστικών με στόχο να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνεκτικότητα, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε να υπάρχει σαφήνεια για τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στον τομέα της ανακύκλωσης σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υλικών που αντιμετωπίζουν, που χρησιμοποιούν. Και η Λίντα Μακάβεν έθεσε ένα ερώτημα για το πώς και πότε θα ξέρουμε περισσότερα για το θέμα της καινοτομία και της αντικατάστασης χημικών ουσιών όταν υπάρχουν εναλλακτικέ δυνατότητες. Υπάρχουν κάποια αρχικά στοιχεία λοιπόν, αλλά είναι πολύ νωρί για να δώσουμε μια απάντηση. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για το κόστος και το όφελος της νομοθεσίας μέχρι τώρα. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να το πράξουμε, αλλά θα συνεχίσουμε το, την εργασία μας για τον τομέα αυτό και δεν μπορώ να σας δώσω τώρα μια συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, αλλά εν καιρό θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Έχουν γίνει ορισμένε μελέτες και έχουν δημοσιευτεί. Ακόμα δεν μπορούμε με μεγάλη εμπιστοσύνη να σας δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Για το τι γίνεται στον τομέα της ε, καινοτομίας και ποια είναι τα ωφέλη τα οποία προσποριζόμαστε σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αυτά ήταν λοιπόν κάποια από τα γενικά ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι αναφέρατε. Υπήρξαν και κάποια λεπτομεριακότερα θέματα τα οποία δεν ξέρω αν θέλετε να σταθούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Θα σταθώ σε ορισμένα από αυτά τα περαιτέρω ερωτήματα τα οποία απευθύνονται στην Κομισιόν. Ο Κρίς Ντέιβις ρώτησε εάν η ελεύθεροι περιορισμή είναι αρκετή διστάζω λίγο να θέσω κάποια συγκεκριμένα όρια για περιορισμούς, γιατί ας δούμε τι κάνει το REACH. Καταχώρηση, διαχειρίζεται τους κινδύνους. Οι εταιρείε έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά αυτό. Υπάρχουν περιορισμοί, περισσότεροι περιορισμοί που δρομολογούνται, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι έχουμε περιοριστεί λοιπόν στους τρεις ε, αυτούς προβλέπεται παρέμβαση των αρχών υποπεριορισμούς φυσικά και επίσης η έγκριση γίνεται πραγματικότητα. Περιμένουμε ότι ανα πάσα στιγμή θα αρχίσει λοιπόν να λειτουργεί. Και όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων των χημικών ουσιών, ε, το REACH είναι το μοναδικό πλαίσιο το οποίο διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους. Δεν βλέπω λοιπόν ε, ένα συγκεκριμένο αριθμό περιορισμών να είναι κατάλληλος από αυτό που ήδη υπάρχει. Σίγουρα, όσον αφορά την επαφή με τις επιχειρήσεις και με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, να σας πω ότι οι συνάδελφοί μου βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με αυτούς και κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να απαντήσουμε στις ανησυχίε και τα ερωτήματά τους. Σίγουρα έχουν πολύ περισσότερα ερωτήματα από ό,τι εμείς. Κάνουμε ό,τι Μπορούμε λοιπόν. Αυτά ήθελα να προσθέσω προς το παρόν. Πιστεύω ότι τα υπόλοιπα ερωτήματα ήταν προς την ΕΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνσε τώρα θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να καλύψω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παρουσίασή μου σε σχέση με την ΕΚΑ. Και φυσικά υπήρχαν ορισμένες ασάφειες σχετικά με τις ε, διάφορες εκπτώσεις ε, στο σύστημα. Η ταυτοποίηση του καθεστώτος σε μία μικρομεσαίας επιχείρησης είναι μια πρόσθετη εργασία την οποία πρέπει να κάνει η ΕΚΑ να διαπιστώσει δηλαδή εάν όντω μια επιχείρηση είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό επιφέρει μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο και είναι κάτι που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν δρομολογείται. Υπάρχει λοιπόν μια αναθεωρημένη πρόταση η οποία επιτρέπει μια έκπτωση 50% μόνο όμως σε περίπτωση όπου μια επιχείρηση στην αρχή της διαδικασίας εξηγήσει με λεπτομέρειες ότι έχει κάνει κάποιο λάθος. Προτού δηλαδή ασχοληθούμε με την επαλήθευση όλων των αποδείξεων, διότι με αυτόν τον τρόπο θα δαπανίσουμε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία στο τέλος θα χρεωθούν σε αυτήν την εταιρεία. Το θέμα λοιπόν είναι σε ποιο σημείο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα μας ενημερώσουν ότι πράγματι έχει γίνει λάθος, δεν είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο. Ταυτόχρονα Εάν όντως έχει διαπιστωθεί αυτό κάτι εγκαίρως, μπορούμε να δεχτούμε εταιρείες που εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι μπορούν να συμπεριληφθούν. Κατ' εξαίρεση είναι αυτό. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τις εταιρείες αυτές. ή να τις επιβαρύνουμε. Διότι μια εταιρεία που δεν θεωρείται μικρομεσαία επιχείρηση δεν είναι κατά ανάγκη τεράστια, μπορεί να είναι στα όρια. Ακόμα και αν μια εταιρεία εξαρτάται κατά το 1 τρίτο από κάποια άλλη μεγαλύτερη, δεν σημαίνει ότι δεν ε, μπορεί να θεωρηθεί μικρομεσία ή όχι. Τώρα, όσον αφορά τις ε, δόσεις που αναφέρατε, δεν προβλέπεται κανονικά από τον κανονισμό κάτι τέτοιο. Ήδη όμως κοιτάζω αυτό αυτή τη στιγμή τις εξαιρέσεις. Εάν δηλαδή κάποια εταιρεία μας ενημερώσει εγκαίρως ότι προτίθεται με να πληρώσει αλλά θα ήθελε να το κάνει αυτό σε δόσεις διότι δεν γίνεται διαφορετικά, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα. Να μην ε, δηλαδή επιβάλλουμε με βάναυσο τρόπο τους κανόνες χωρίς καμία εξαίρεση, αλλά εάν υπάρχει πραγματικά καλή αιτιολόγηση να κοιτάξουμε για εξαιρεσει. Το ίδιο και με ανάκληση καταχωρήσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, έχει ανακληθεί δηλαδή ο αριθμός καταχώρησης μιας εταιρείας και έχουν παρατηρηθεί στην περίπτωση αυτή λάθος πρακτικές εξαγορά μιας εταιρείας από κάποια άλλη. Εδώ χρειάζεται λεπτομερέστατη ταυτοποίηση και επαλήθευση στοιχείων. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι κανόνες με τους οποίους μπορεί να είμαστε σχετικά ευέλικτοι, να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε ορισμένε εταιρείε εντός λογικών ορίων πάντοτε να μας παρουσιάσουν δικαιολογητικά, τα οποία θα επιτρέψουν μια ενδεχόμενη εξαίρεση από τους κανόνες. Τώρα, όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα, να σας πω ότι εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε μαζί με το GRC και έχουμε εγκρίνει ορισμένε εναλλακτικές μεθόδους για τις δοκιμές σε ζώα προτού τις οριστικές προθεσμίες σε περιπτώσεις που απαιτούνται δοκιμές σε ζώα. Και πραγματικά προσπαθούμε μαζί με τους συνεργάτες μας και με την ερευνητική κοινότητα να βρούμε αυτές τις εναλλακτικέ, να τις εγκρίνουμε και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τις δεχτούμε και να συμπεριληφθούν στα παραρτήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν καλές προοπτικές για θετική εξέλιξη. Όσον αφορά τώρα τους περιορισμούς, νομίζω πως τους κάλυψα. Επίσης για τη δημοσίευση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Να σας πω ότι με το να διαγράψουμε το όνομα μιας εταιρείας δεν σημαίνει τίποτα. Τη στιγμή που δημοσιεύσουμε εμείς κάτι, μπορεί η εταιρεία αυτή να έχει ήδη συμμορφωθεί με τις απαιτήσει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δημοσιοποιήσουμε το όνομα μιας εταιρείας εάν ήδη έχει διορθώσει τα σφαλματά της. Διότι αυτό που θέλουμε σε τελική ανάλυση είναι να ενημερώνονται τακτικά οι φάκελοι στα μικρόα καταχώρησης προτού χρειαστούν ρυθμιστικές δράσεις. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθούμε να ρυθμίσουμε την ποιότητα των φακέλων αυτών. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να μην δημοσιεύονται τα ονόματα λοιπόν των εταιρείων αυτών. Δεν είναι δύσκολο, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, να μάθει το όνομα μιας ε, τέτοιας εταιρείας. Υπάρχουν διάφοροι στότοποι και υπάρχουν και έμεση τρόποι για να μάθει κανείς ποιες εταιρείες έχουν σχέση με ποια ουσία. Το κύριο Μητρό λοιπόν είναι υπεύθυνο. Αλλά η εταιρεία που είναι υπεύθυνη πολλές φορές ενεργεί εκπροσωπώντας και άλλες μικρότερες. Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει σε σχέση με την ποιότητα των δεδομένων και αυτό θα το έχω λοιπόν στην παρουσίασή μου στη συνέχεια αλλά προς το παρόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά τερματικά σημεία αν θέλετε μέσω ε, ελέγχων στοχευμένων για τη συμμόρφωση και θα καταλήξουμε σε πολλές αποφάσεις για τα θέματα αυτά και όπως είπε και ο άλλον. Μπορεί οι εταιρείε χωρίς ε, επαρκή ε, εμπειρογνωμοσύνη σε επιστημονικό επίπεδο <clears throat> δεν έχουν προβεί σε ένα κανονικό σε μια κανονική δοκιμασία. Θα τους δώσουμε την ευκαιρία λοιπόν να μετανοήσουν και να βελτιώσουν την αντιμετώπιση τους. Δεν, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να δικαιολογήσουμε αν δεν χρειάζεται μια δοκιμασία και αν έχουν άλλες <clears throat> πληροφορίες και άλλους τρόπους να παρουσιάσουν δεδομένα για το VVBT, για το PPTPT. Αυτά λοιπόν. Μπορώ να κάνω τώρα την ε, ομιλία μου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είναι μια μεγάλη ε, τιμή για μένα να μπορώ να ανατρέξω στα πρώτα πέντε χρόνια του Ρίτσου. Στα επόμενα 10 λεπτά θα σας παρουσιάσω ορισμένα ιστορικά στοιχεία και θα σας τονίσω και ποιες είναι οι βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν σε σχέση με το REACH και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Φάρμακα. Και φυσικά νομίζω ότι ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανταλλαγές απόψεων. Πολλοί από εσά θυμόσαστε ότι το πότε εγκρίθηκε το REACH και εγώ το θυμάμαι, αλλά δεν ήξερα τι περίμενε για τι είχε για μένα η μοίρα να πάω στο Ελσίνσκι να δημιουργήσω την, ε, τον Ευρωπαϊκό Φορέα Χημικών Ουσιών και να προσπαθήσω να καλύψω τις νομοθετικές επιταγές για αυτόν τον οργανισμό. Αυτά τα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα και τα πιο εξαντλητικά της επαγγελματικής μου ζωής. Και εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου στην ΕΚΑ ικανοποιούνται ιδιαίτερα για τον κέριο ρόλο που διαδραματίσαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο ασφαλή και πιο υγιή. Πολλοί από εσά και οι προκάτοχοι σας σε αυτή την Επιτροπή σίγουρα μπορούν να συμμεριστούν την ε, περηφάνεια που νιώθουμε όλοι μας και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη που πήρε η ΕΚΑ όλα αυτά τα χρόνια από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το ΡΙΤΣ είναι μια συλλογική προσπάθεια <clears throat> και νομίζω ότι έχουμε καταδείξει την ικανότητά μας να εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου. Επίσης γνωρίζω ότι στην αρχή του δρόμου πολλοί από εμά περιμένανε να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, αλλά είχαν και φόβους ότι θα γίνει το χειρότερο, όπως είπε και ο Κρίς λόγω της τεράστιας κλίμακος των προκλήσεων που είχαν ενώπιόν μας και του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος. Όπως όμως έχει δείξει και η πρόσφατη επισκόψη για το ΡΙΤΣ από την Κομισιόν, παρά όλες αυτές τις προκλήσεις το ΡΙΤΣ λειτουργεί πολύ καλά και η ΕΚΑ έχει καταφέρει να παίξει το ρόλο. Σας θυμηθούμε ποιε ήταν αυτές οι προκλήσεις. Η αναστροφή του βάρους αποδείξεως, οι πιέσει προ τη βιομηχανία για να συνεργαστεί μαζί μα, οι νέοι τρόποι λειτουργία για τι αρμόδιε αρχέ και η ταχύτητα, <clears throat> η επιτάχυνση της λήψης μέτρων για τη διαχείριση του κινδύνου, η ανάγκη να δημοσιεύσουμε στοιχεία για όλα, όλες τις χημικές ουσίες στο διαδίκτυο και η ανάγκη να έχουμε βελτιωμένη πληροφόρηση ασφάλειας για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τους ε, καταναλωτές, ενώ αποφεύγοντας τη δοκιμασία σε σώα. Σήμερα στην ε, ιστοσελίδα της ΕΚΑ μπορείτε να βρείτε στοιχεία από πάνω από 33.000 φακέλους για πάνω από 8.000 ουσίες που είναι στην αγορά στην Ευρώπη. Οι περισσότερε από αυτέ τι πληροφορίε δεν υπήρχαν πριν από τώρα και τώρα έχουν συγκεντρωθεί και είναι διαθέσιμε σε όλου του ενδιαφερόμενου. Έχουμε επίση 138 ουσίε που είναι πολύ ανησυχητικέ στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών και 22 ουσίε στον κατάλογο έγκρισης και εργαζόμαστε προ το στόχο του 2020 <coughs> που είναι το να έχουμε όλες αυτές τις ουσίες που είναι, χαρακτηρίζονται ως SVHC στον κατάλογο. Σήμερα ο συνδυασμός των επιταγών για αυτούς που καταγράφουν ουσίες και για τους χρήστες τους συμβάλλει σε μια πιο ε, ασφαλή χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών και αντικατάσταση των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών είτε μέσα από ρυθμιστική δράση είτε προορατικά. Θα γίνει όλο και περισσότερη αντικατάσταση αυτών των ουσιών, κάτι το οποίο είναι σημαντικό στόχο για το ΡΙΤΣ. Όπω ξέρετε, σήμερα ε, επίκειται το επόμενο ορόσημο τη ΡΙΤΣ, η δεύτερη καταληκτική ημερομηνία για την καταγραφή ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε όγκους μεταξύ 100 και 1000 τόνων το χρόνο. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό μου στο Ελσίνκι διεκπεραιώνει χιλιάδες νέους φακέλους στις τελευταίες μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία. πλησιάζουν και οι τελευταίες μέρες για την καταγραφή όπως ξέρετε. Η ΕΚΑ θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα την επόμενη Δευτέρα εδώ στις Βρυξέλλες και θα παρουσιαστεί στο διαδίκτυο η συνέντευξη τύπου ώστε να μπορέσετε από μόνοι σας να παρακολουθήσετε τα αποτελέσματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά σε σχέση με μια τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Βέβαια δεν είναι όλα ροδόχρωα σε ό,τι αφορά την ιστορία του Ρίτς και θα σας υπενθυμίσω τέσσερις τομείς όπου μπορούν να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις για την ΕΚΑ. Πρώτα απ' όλα η ποιότητα των στοιχείων που παρουσιάζονται στους πακέλους καταγραφής, η πληροφορία για τις χημικές ουσίες και η πληροφορία για το πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά και ασφαλώς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ΡΙΤΣ. Με, όταν έχουμε στοιχεία υψηλής ποιότητας τα οποία δίνονται στους χρήστες μπορούν να υπάρχουν μέτρα εξασφάλισης και να χρησιμοποιηθούν οι ουσίες αυτές με ασφαλή τρόπο. Χωρί όλα αυτά τα στοιχεία δεν θα μπορούσαν να αντίσουν χίλια λουλούδια. Η ΕΚΑ προσπαθεί να βοηθήσει με το να δείχνει πώ θα πρέπει να είναι οι φάκελοι, ποια θα είναι η κατάλληλη πρακτική βοήθεια, η μεταλαμπάδευση καλύτερων πρακτικών και μια ετήσια αξιολόγηση θα εξετάζουμε τουλάχιστον τα 5% των φακέλων και θα εξετάζουμε στοχευμένα ορισμένους άλλους τομείς χημικών ουσιών. Αλλά τελικά είναι οι εταιρείε οι οποίες θα πρέπει να βελτιώσουν και να ε, ενημερώσουν τους φακέλους τους το ταχύτερο δυνατό προτού τους υποχρεώσουμε να το κάνουμε αυτό. Ένας δεύτερος τομέας βελτίωσης που θα βοηθήσει την έκανε πτήξη να επιτύχει το στόχο του ΡΙΣ είναι να βοηθήσουμε τις τεχνολογικές και επιστημονικές ε, εξελίξεις όπως είναι η νανοτεχνολογία και η αντιμετώπιση των ενδοκρινικών διατρακτών. Η νανοτεχνολογία δεν παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή σε μεγάλο επίπεδο στους φακέλους. Είναι πολύ λίγοι φάκελοι που αναφέρουν αυτές τις ουσίες. Γι' αυτό, επειδή και το Ρίτσα αναφέρεται επακριβώς στους, στις νανοουσίες, Πολλέ εταιρείε δεν τι περιλαμβάνουν στους φακέλου του. Αλλά η εμπειρία των ΗΠΑ καταδεικνύει ότι οι νέε ουσίε έχουν ένα υψηλό ποσοστό ουσιών που βρισκόνται σε νανομορφή. Γι' αυτό περιμένουμε την ε, αναθεώρηση των παρατημάτων του ΡΙΤΣ από την Κομισιόν για να μπορέσουμε να καλύψουμε και ουσίε οι οποίε βρίσκονται σε νανομορφή πρωτού αναπτύξουμε περαιτέρω κατευθυντήρε γραμμέ και βοήθεια προ τι εταιρείε που θα του επιτρέψουν να τι καταγράφουν με τον κατάλληλο τρόπο και να ενημερώνουν του φακέλου του όταν αυτό είναι απαραίτητο και να έχουμε την κατάλληλη κατεύθυνση για τη διαχείριση κινδύνου. Το ίδιο ισχύει και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, όπου περιμένουμε και από την Κομισιόν να περατώσει και να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της για τα κριτήρια εντοπισμού αυτής της τόσο σημαντικής ομάδος <clears throat> ουσιών που οδηγούν σε υψηλή ανησυχία. Τρίτο θέμα είναι η αναθεώρηση από την Κομισιόν των Πληροφοριών που χρειάζονται για οι ουσίες που έχουν παραγωγή ή εισαγωγή μεταξύ ενός και τόνων. Φυσικά θα μπορούσε να υπάρχει νανοπαραγωγή σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγή, όπου είναι περιορισμένε οι υποχρεώσει, παροχή πληροφοριών και δεν υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει μια ε, έκθεση για την χημική ασφάλεια. Ελπίζουμε ότι το έργο τη Κομισιόν πέρσι του χρόνου θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτά τα θέματα. Τέλο. συμφωνούμε με την Κομισιόν, θα πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξη που δίνουμε στι μικρότερε εταιρείε. Οι μεγάλες χημικές <clears throat> εταιρείες στην Ευρώπη είναι πεπισμένες ότι τα ωφέλη του ρίτς είναι υπέρτερα του κόστους. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις πιο μικρές επιχειρήσεις. Οι προτάσεις μου έχουν σε στόχο να αλλάξουν τον αρνητικό αντίκτυπο και την αρνητική αντίληψη του ρίτς από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εμπειρία όλο και περισσότερο μας δείχνει ότι το ποσοστό των μικρότερων εταιρεών που καταγράφονται μέσα σε αυτή την περίοδο για την καταληκτική προθεσμία είναι περίπου το ίδιο, δηλαδή περίπου 20% του συνόλου μαζί με όλους τους εμπλεκομένους. Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να πλησιάσουμε τις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι προμηθευτές, είτε δημιουργούν χημικές ενώσεις, είτε είναι επαγγελματικοί χρήστες, παραγωγή κτλ. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν ακόμα για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους ή το πώς να εκμεταλλευτούν καλύτερα το ρίτσο. Μια πιο στοχευμένη αντίληψη είναι απαραίτητη και σχετικές εκστρατείες θα πρέπει να γίνουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές και οι μικρότερε εταιρείε θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμορφωθούν απόλυτα με το ΡΙΖΟ. Θα πρέπει να καταλάβουν ποιε είναι οι χημικέ ουσίε που παράγουν και χρησιμοποιούν και να δώσουν πληροφορίε για το πώ να τι χρησιμοποιήσουμε με πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Συγχρόνω όμω είμαστε έτοιμοι να τι βοηθήσουμε να συμμορφωθούμε. Με, έχουμε ένα πολύ θετικό ιστορικό προ την κατεύθυνση αυτή μαζί με τα εθνικά γραφεία βοήθεια για να δίνουμε υποστήριξη και βοήθεια σε όλες τις εθνικές γλώσσες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η γλώσσα να μην αποτελεί ένα εμπόδιο. Επίσης, συζητάμε με τους διαπιστευμένους ε, εμπλεκόμενους τις μορφές πρόσθετης βοήθειας που μπορούμε να δώσουμε. Θέλουμε επίσης να δούμε τι μεγάλες εταιρείε να βοηθούν τις μικρές εταιρείε με δική του πρωτοβουλία. Οι εμπειρογνώμονε τουρίστε σε μεγάλες εταιρείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να πληροφορούν τις μικρότερες εταιρείες όπως γίνεται εδώ στο Βέλιο και έτσι οι, οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος πρόσβαση δεδομένων για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όπω βλέπετε, η αξιολόγηση τη ΕΚΑ για τι απαραίτητε βελτιώσει στο σύστημα REACH συμφωνούν με την ε, επισκόπηση και αναθεώρηση τη Κομισιόν λόγω των πολλών συστάσεων που υπάρχουν σε σχέση με την συμμετοχή της ΕΚΑ, έχουμε αποφασίσει να ενσωματώσουμε αυτές τις ανάγκες στο επόμενο στρατηγικό πολιτές πρόγραμμα εργασίας για το 2014-2018 της ΕΚΑ. Το έγγραφο αυτό είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας για δημόσια διαβούλευση και ένα τελικό κείμενο <clears throat> θα εγκριθεί από, την, από το Διοικητικό μας Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο. Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής, Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ευκαιρία να είμαι εδώ ενώπιον σας σήμερα και να σας αναφέρω τις σκέψεις μου με την αναδρομή αυτή στα πρώτα πέντε χρόνια του ΡΙΤΣ. Πιστεύω ότι σε, στα επόμενα πέντε χρόνια, μετά από πέντε χρόνια, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούν να σας πληροφορήσουν μαζί με τον διάδοχό μου στην ΕΚΑ για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και μεγαλύτερη θετική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον μέσα στα πλαίσια αυτού του θαυμάσιου εγχειρήματος του Ριτς. Ευχαριστούμε πολύ Γκέρτ. Περνάμε τώρα στον δεύτερο κύκλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους εσάς, εσάς και την ομάδα σας στο Ριτς, που τα τελευταία πέντε χρόνια είστε ένα οχυρό που προφυλάσσει όλους εμάς. Πρέπει πραγματικά να είμαστε περήφανοι για αυτά που έχετε καταφέρει στα πέντε χρόνια λειτουργία σας όσον αφορά την ενομοθεσία για τις χημικές ουσίες παρά τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί παρά το φορτωμένο σας πρόγραμμα και τον λίγο χρόνο. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και όλοι σας την ομάδα στο Ελσίνκι. Αρχίζουμε τώρα τη συζήτηση. Will Pog, Corinne Lepage και Chris Davis. Pavel Pog. Με ναι, μια πολύ σύντομη ερώτηση μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα μας διανεμηθούν τα στοιχεία. Σίγουρα, λέει πρόεδρος. Μπορούμε να το κάνουμε. Pavel Ποκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τρία πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή. Αναφέρατε τους στόχους για μη τοξικό περιβάλλον, περιβάλλον χωρίς τοξίνες. Πιστεύω πως αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί μόνο σε διεθνές επίπεδο. Και φυσικά το REACH δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις και επιπλοκέ στις ενές χώρες που συμμετέχουν. Θέλω να ρωτήσω, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το REACH βοηθάει ή δεν βοηθάει στη δημιουργία πολιτικών διαχείρισης χημικών ουσιών και αποβλήτων. Έπειτα, όσον αφορά την πληροφόρηση, πιστεύετε πως η διάδοση των πληροφοριών από την ΕΚΑ στους πολίτες έχει αποτελέσματα, είναι λειτουργική, είναι χρήσιμη όσο πρέπει. Ή πιστεύετε ότι ακόμα υπάρχουν κοινά, κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και τελευταία ερώτηση πάλι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω πως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες δεν μπορούν ε, να ελεγχθούν επαρκώς και οι επιπτώσεις τους είναι και συγκεντρωτικές επίσης. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, Πάβαλ. Κορίν Λεπάζ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είχα δύο ερωτήσεις να σας θέσω. Εν μέρη απαντήσατε στην μία που αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που όπως είπατε δεν μπορούν να ελεγχθούν ακόμα στο πλαίσιο του ΡΙΤΣ καταλήλως. Ε, πέρα από τη λεπτομερή αναφορά και τη στρατηγική αεροπλούς, η επόμενη λειτουργία στην οποία θα ελέγχονται οι ενδοκρινικοί διαταράκτες μέσα στη διαδικασία διοδότησης του ΡΙΤΣ είναι να ελεγχθούν ε, όντως οι διακοιμάνσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών μέσω πιο βέβαιων εναλλακτικών. Ε, επίσης και για τα βιο ε, ανθεκτικά, σωρευτικά χημικά στοιχεία, Η ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η δεύτερη αρχή αφορά το θέμα της υποκατάστασης η υπηρεσία σας, ο οργανισμός σας, κύριε Διευθυντά, έχει να παίξει ρόλο κλειδί στην προώθηση και στην εφαρμογή αυτής της αρχής. Ο κανονισμός REACH ενθαρρύνει την υποκατάσταση, αλλά ο οργανισμός σας έχει παίξει ουσιαστικότατο ρόλο. Πιστεύετε πως μπορείτε ακόμα να ενδυναμώσετε αυτό το ρόλο στα επόμενα χρόνια. Και τελευταία παρατήρηση για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι πολύ σημαντικό οι βασικές αρχές του κανονισμού REACH, ε, ε, όπως η αρχή της πρόληψης και της υποκατάστασης, να εφαρμοστούν σωστά. Μπορούμε να βελτιώσουμε περισσότερο την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σαν το χάσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Ντάνσετ για την παρουσίασή του. Μετά τον πρώτο γύρο είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις και περίμενα απαντήσεις σε αυτές. Στην παρουσίαση του κυρίου Ντάνσετ. Αλλά νιώθω πως δεν έλαβα τις απαντήσεις που ήθελα. Όσον αφορά τους ε, αριθμούς καταχώρησης, μας είπατε ότι το σκέφτεστε, σε περίπτωση που ο φάκελος συνεχίζει να μη συμμορφώνεται παρά τις επιστολές που θα έχετε στείλει μετά από τον πρώτο έλεγχο. Και αφού διαπιστωθεί ότι ο φάκελος δεν συμμορφώνεται και αφού έχετε ζητήσει από την εταιρεία να διορθώσει το πρόβλημα αυτό. Έχετε αφαιρέσει τον αριθμό καταχώρησης λοιπόν μέχρι τώρα. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίες για τα CMR και τα PBT, ούτε εδώ πιστεύω πως έλαβα κάποια απάντηση στις ερωτήσεις μου. Ποια είναι τα σχέδιά σας. Τι σκοπεύετε να κάνετε όταν διαπιστώνετε ότι μόνο 20% των φακέλων περιέχουν πληροφορίες για το εάν οι ουσίες είναι, ανήκουν στο CMR ή στο PBT. Και το 80% του περιεχομένου δεν παρέχει τέτοιες πληροφορίες. Θα ήθελα να ξέρω πόσες ουσίες είναι αυτές και τι κάνετε έτσι ώστε να έχετε αυτές τις πληροφορίες από τις εταιρείες και πότε τις έχετε. Και όσον αφορά τα νανοηλικά, μας είπατε ότι περιμένετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να γίνουν αλλαγές στα παραρτήματα του REACH έτσι ώστε να βελτιωθεί το σύστημα για τα νανοηλικά. Για την αξιολόγηση όμως του κινδύνου χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με αυτόν και πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στις ουσίες αυτές. Οι πληροφορίες όμως αυτές σχετικά με την έκθεση λαμβάνονται μόνο από τις εκθέσεις ε, ασφαλείας των χημικών ουσιών, οι οποίες προς το παρόν απαιτούνται μόνο από χημικές ουσίες οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των πάνω από 10 τόνους, όχι για μικρότερες ποσότητες χημικών ουσιών. Ούτε για τα CMR. Μέχρι τώρα σχεδόν καμία από τις χημικές ουσίες που είναι καταχωρημένη ως νανοουσία υπόκειται σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Και κάτι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο έχει συντάξει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, στην οποία αναφέρεται ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένη νομοθεσία για τα νανοηλικά. Όχι μόνο το να αλλάξουμε τα παραρτήματα, δεν ε- επαρκεί αυτό. Το πρόβλημα θα συνεχιστεί δηλαδή ότι δεν θα λαμβάνουμε καμία πληροφορία σχετικά με την έκθεση αυτές τις ουσίες, οι οποίες πληροφορίες περιέχονται μόνο στις εκθέσεις ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και... Ευχαριστώ πολύ Σάτου. Έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των ομιλητών και σας ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, που μου απευθύνθηκαν, που μου υποβλήθηκαν. Για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες έχουμε ήδη εντοπίσει κάποιες ουσίες ως ενδοκρινικούς διαταράκτες παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ε, ε, καθιερωμένα ευρωπαϊκά κριτήρια, ενωσιακά μάλλον κριτήρια, ε, υπάρχουν ε, ενδείξεις ή αποδείξεις ε, ώστε να μπορεί κανείς να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα ότι δηλαδή αυτές οι ουσίες έχουν αυτές τις ιδιότητες και τις έχουμε τοποθετήσει στο κατάλογο και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε μάλιστα τη δυνατότητα να τις περάσουμε και στο κατάλογο αδειοδότησης. Όμως κατά τη γνώμη μου είναι αλήθεια ότι για να καθοριστούν οι διαταράκτες θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύνολο σαφών κριτηρίων για τον ορισμό τους. Το ρόλο, ο ρόλος της υποκατάστασης τώρα. Φυσικά έχουμε, προωθούμε την υποκατάσταση ήδη σε μεγάλο βαθμό μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης. Και αυτό επειδή έχει αποδειχτεί για παράδειγμα ότι για τις πρώτες ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο έγκρισης ε, αδειοδότησης όπου η προθεσμία έχει ήδη περάσει για την αίτηση αδειοδότησης δεν υπήρξε καμία αίτηση. Κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον να χρησιμοποιήσει αυτές τις ουσίες, σημαίνει αυτό. Οπότε, ε, θα έπρεπε επίσης να αναμένετε ότι στο μέλλον εν γέννη θα έχουμε λιγότερα λιγότερες αιτήσει για διοδότηση από ό,τι αρχικά είχε εκτιμήσει η Κομισιόν. Και αυτό είναι απόδειξη της επίπτωσης που έχει ο, ε, ε, καταχώρηση στον κατάλογο των χημικών αυτών ουσιών. Επίσης έχουμε σχέδιο να προαναπτύξουμε στο site μας πώς μπορεί αυτό να κινητοποιήσει την υποκατάσταση. Και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ε, από τη στιγμή που υπάρχει η, ε, ο κατάλογος των ε, αδειοδοτήσεων θα παίξει αυτό ρόλο. Σήμερα λάβαμε, ε, αυτή την εβδομάδα λάβαμε την πρώτη αίτηση για αδειοδότηση. Θα δούμε λοιπόν ποιε είναι οι δυνατότητε υποκατάσταση για το συγκεκριμένο χημικό, στη συγκεκριμένη χημική ουσία. Είναι πλέον δηλαδή θέμα χρόνου ώστε αυτή η διαδικασία που θέλατε να έχετε οπωσδήποτε θα δείξει πια τις πρακτικές της επιπτώσεις. Και ένα ερώτημα για την κυρία Χάση. Δεν θέλω να μην απαντήσω στο ερώτημά σας. Θέλω απλά να διαποσαφηνίσω για μια ακόμη φορά αυτό που ήθελα να πω όσον αφορά την απόσυρση των ε, αριθμών καταχώρησης. Ναι, έχουμε ήδη αποσύρει κάποιους αριθμούς καταχώρησης, αλλά αυτό είχε περισσότερο να κάνει με την επαλήθευση SME. Για να αποσυρθεί ένας αριθμός καταχώρησης από μια εταιρεία που δεν συμμορφούνται, υπάρχει όχι μόνο το στοιχείο ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει συμμορφωθεί προς την τελική απόφαση, αλλά επίσης υπάρχει και ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν να μπορέσουμε να ξαναδούμε ε, το θέμα. Και αυτό είναι οι αρχές επιβολής πρέπει να ενεργήσουν πρώτες για την μη συμμόρφωση. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις εκδίδουμε ε, μια επιστολή μη συμμόρφωσης και ζητούμε από τις αρχές επιβολής να παρέμβουν. Αυτό προβλέπει το ΡΙΤΣ σύμφωνα με την ερμηνεία της νομοθεσίας. Και μετά μπορούμε να ξαναδούμε το ντοσχέ. Επίσης, δεν σημαίνει ότι υπό οποιοδήποτε μορφή μη συμμόρφωσης μπορούμε να αποσύρουμε τον αριθμό καταχώρησης. Ε, πρέπει να είναι μια σοβαρή ε, πτυχή που να ενοχλεί την σωστή διαχείριση των χημικών ουσιών. Τα, σε σχέση τώρα με τα C-Market PBTs, στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται στο βασικό ντοσιέ, γιατί και εκεί πρέπει να υπάρχει ταξινόμηση. Είναι μια κοινή πτυχή των ε, κοινών αν δούμε λοιπόν το... θα, δούμε, θα, θα δούμε την ταξινόμηση του ομίλου ή της ομάδας εταιριών που έχουν καταχωρήσει το προϊόν. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες εταιρείες που πουλούν αυτά τα προϊόντα ε, σε μεγάλες ποσότητες και μπορεί να έχουν κοινοποιήσει σε διαφορετική ταξινόμηση. σύμφωνα με το CLP και εκεί έχουμε μια βάση CLP, μια πλατφόρμα CLP όπου οι εταιρείε πρέπει να συζητούν αυτές τις διαφορές σε ταξινόμησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, πώς θέλουμε να συμπληρώσουμε το κενό της ενημέρωσης. Ο μόνος τρόπος είναι εξετάζοντας τις σημαντικές, τα σημαντικά σημεία εισόδου για το κατά πόσο ε, μια ουσία είναι CMI ή PBD ή οτιδήποτε άλλο. Και ε, έτσι εξετάζουμε τη συμμόρφωση όλων των ντοσιέ. Ταυτόχρονα και μετά πάμε σημείο προς σημείο για να εντοπίσουμε ποια ντοσιέ έχουν μειονεκτήματα και μετά εκφέρουμε, λαμβάνουμε μάλλον αποφάσεις. Αυτό κάνουμε. Τα άλλα ερωτήματα νομίζω απευθύνονταν στην Επιτροπή. Η Κομισιόν λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για, τις, για τα νανοηλικά όπως ανέφερε η Σάτου Χάση έθεσε το ερώτημα του αν χρειαζόμαστε πρόσθετους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε τα νανοηλικά η μεταρρύθμιση του κανονισμού από τα παρατήματα. Απλώς θέλω να πω ότι τον Ιούλιο ξεκινάμε μια δημόσια διαβούλευση πολύ σύντομα δηλαδή για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα νανοηλικά για να υπάρξει και μεγαλύτερη σαφήνεια. Και να εξασφαλίσουμε και πιο ασφαλή χρήση. <clears throat> Με τη δημόσια αυτή διαβούλευση και, την, και τον έλεγχο αντικτύπου θα προχωρήσουμε. Αλλά το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αν θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο για να κάνουμε κάτι στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τη βάση των διατάξεων που το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο έχουν ήδη εγκρίνει σε ό,τι αφορά τις ε, εκτελεστικές διατάξεις. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν περισσότερο το πώς θα καταλήξουμε σε αποτελέσματα και γι' αυτό δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ρυθμιστική ανασφάλεια με το να ανοίξουμε και πάλι το θέμα αυτό. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία του Κοινοβουλίου και το εξετάσουμε αυτό μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου αντικτύπου και διαβούλευσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Είπε και ο Ντάνσετ ότι είναι απαραίτητο να έχουμε σαφέστερα κριτήρια για την ε, αναγνώριση των ενδοκρινικών διαταρακτών Κάναμε μια μεγάλη διεθνή συνδιάσκεψη πέρσι και έχουμε μια στρατηγική η οποία είναι ίσως πεπαλαιωμένη και προσπαθούμε να δούμε τι καινούριο μπορούμε να προτείνουμε μέσα στα πλαίσια μιας νέας στρατηγικής για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε στο άμεσο μέλλον για κριτήρια εντοπισμού και αναγνώρισης αυτών των διαταρακτών. Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη μέσα στο ΡΙΤΣ για την διεύρυνση των διατάξεων σε σχέση με ουσίες που είναι υψηλής ανησυχίας λόγω του ενδοκρινικά διαταρακτικού χαρακτήρα τους και θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση αυτή την επόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, για όλα αυτά τα νέα κριτήρια που πρέπει να ακολουθηθούν. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ε, υποκατάσταση όλων αυτών των ουσιών, την αντικατάστασή τους να από πιο ασφαλείς ουσίες και ρώτησε η Λίντα Μακάβεν προηγουμένως για το τι μπορούμε να κάνουμε στα θέματα αυτά. Έχουμε δεσμευτεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 να παρουσιάσουμε τα πιο καινοτόμα στοιχεία αυτής της στρατηγικής. Και οι άλλες χώρες τι κάνουμε με αυτό το ερώτημα είναι φανερό ότι πολλές χώρες που παράγουν χημικές ουσίες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ελβετία ήταν πάρα πολύ αμυντική στην αρχή μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Αλλά η συζήτηση έχει οριμάσει, η ελβετική κυβέρνηση εξετάζει αν θέλει να ενταχθεί πλήρως στο σύστημα του ΡΙΤΣ, αλλά ακόμα αμφιταλαντεύεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε μια εκβάθρον αναθεώρηση της νομοθεσίας τους για τις χημικές ουσίες, να δουν τι μπορούν να κάνουν στη δική τους αγορά, που δεν βέβαια εμπνέεται πλήρως από το αλλά έχει παρόμοιους στόχους όπως το ΡΙΣ, δηλαδή να αντιμετωπίσει την, τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Υπάρχει λοιπόν και κάποια κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο για τα θέματα αυτά. Για την πληροφόρηση των πολιτών μέσα στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης. Ακούσαμε τις απόψεις των εμπλεκομένων και γενικά πιστεύουν ότι πήγαινε πολύ καλά ο φορέας για το ΡΙΣ σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών. Και πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν και περαιτέρω Ανταλλαγέ πληροφοριών με τις, μεταξύ των εταιριών και της Κομισιόν, βέβαια υπό την προϋπόθεση της εμπιστευτικότητας, που είναι σαφές αυτό. Η Σα του Χάση είπε, γιατί το 2020, γιατί να περιμένουμε τόσο πολύ. Η δική μου απάντηση είναι γιατί ο αντιπρόεδρο Ταγιάννη και ο επίτροπο Ποτόσνικ θεώρησαν την απαραίτητο να έχουμε ένα οδικό χάρτη. Μεγάλη πρόοδο έχουμε επιτύχει, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε και ένα οδικό ε, χάρτη. Μέσα στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε να καταγράψουμε τις 130 επικίνδυνες ουσίες μέχρι το τέλος του χρόνου και θεσπίζουμε και στόχους για το περαιτέρω Γι' αυτό είναι απαραίτητο να θεσπίσουμε ένα ενδιάμεσο στόχο σε αυτό τον οδικό χάρτη, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κάλυψε τα πάντα εκτός από δύο σημεία. Οπότε θα απαντήσω σε αυτά την κυρία Λεπάζε. Ρωτήσατε γιατί η, αν και κατά πόσο η αρχή της πρόληψης και της υποκατάστασης αντικατοπτρίζονται και εφαρμόζονται επαρκώς. Νομίζω πως ναι. Και έπειτα υπήρχε μια πιο ειδική ερώτηση σε σχέση με την ε, αδειοδότηση των PBTs και των ενδοκρινικών διαταρακτών. Νομίζω αυτό αναφέρεται ε, μέσα στο ε, στον κανονισμό για το αν υπάρχουν εναλλακτικέ ή ε, ε, εφικτές λύσεις. Ναι, φυσικά. Αυτό ακριβώς λέει ο κανονισμός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας θα ήθελα να δώσω το λόγο στο δικό μας εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρώην Ευρωβουλευτή Άλεν Λαπαρεούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ κυρίως που με καλέσατε ε, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για την νομοθεσία Ρίτς. Ένας ε, προβληματισμός που ίσως να ανήκει στο όνειρο και στο, σε έναν ιδανικό κόσμο, αλλά θα ξέρετε ότι ο οργανισμός αυτός εργάστηκε με πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση, όπως επιστώσετε και στην έκθεσή μου, αλλά και εσωτερικά έθεσε έναν στόχο, δηλαδή ο οργανισμός αυτός να αποτελέσει παγκόσμια αναφορά για την γνώση στα χημικά προϊόντα. Διερωτώ λοιπόν αν τα Κάτι μελη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν επίσης να υιοθετήσουν αυτό το στόχο, δηλαδή ο οργανισμός αυτός να είναι παγκόσμιος οργανισμός για τα χημικά, αλλά και το ΡΙΤΣ να αποτελέσει ένα κανονισμό παγκόσμιας εμβέλειας για τα χημικά προϊόντα. Ο Χέλμουντ Σμιτ, παλιός καγκελάριος της Γερμανίας, είπε ότι... Ποιος έχει οράματα να πάει να δει το γιατρό. Αυτά θα αποκλίνοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σας δουλειά. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετέχους. Στην αρχή της θητείας μου εδώ στο Κοινοβούλιο είχα ασχοληθεί με το REACH και πιστεύω ότι από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει τρομερά βήματα προς τα εμπρό. Το REACH πραγματικά είναι επιτυχές, δεν πρέπει όμως να το παραμελήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά και να διασφαλίσουμε την συγχρηματοδότηση. Η νομοθεσία κοστίζει και μια καλή νομοθεσία πρέπει να έχει σοβαρή χρηματοδότηση. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είμαστε, να κάνουμε τσιγκουνιές. Αυτά θα ήθελα να αποκλίνοντα. Ευχαριστώ όλους. Καλό ταξίδι σας εύχομαι σε όσους από εσάς γυρίζετε σήμερα στο σπίτι σας. Καλό μεσημέρι. Σας παρακαλώ να είστε όλοι στην ώρα σας εδώ. Στις 3 ακριβώς θα αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Έχουμε τεράστια ψηφοφορία. Να φέρετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, παρακαλώ και δεν θα είμαι καθόλου επίοικη σε όσους αργήσουν. Γεια σας.